Buenas Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών. Θα μου επιτρέψετε όμως προηγουμένως, πριν περάσουμε στα ουσιαστικά σημεία, να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτον, η κυρία Ματσόνη, η Προεδρός μας, δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα την αντικαταστήσω λοιπόν εγώ για σήμερα. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι θα έχουμε σήμερα μεταξύ μας μία αντιπροσωπεία. Μου γράφει εδώ, κάπου μου το έχει βάλει το γραμματεία να το διαβάσω. Λοιπόν, είναι μια αντιπροσωπεία από την Σαξονία. Ομάδα εργασίας συγκεκριμένα από την Επιτροπή Αναφορών η Τσεντεού ουσιαστικά, είναι αντιψώλη της Τσεντεού. Χανερόλ Ντίσχολτα είναι η επικεφαλή επτά μέλη απαρτίζουν την προσωπία, είναι πίσω στο βάθος της αίθουσα. Και φυσικά τους καλωσορίζουμε θερμά. Ο κύριος Γιάρ έπρεπε να είναι εδώ, αλλά επειδή έρχονταν από τη Γερμανία καθυστέρησε και θα έρθει λίγο αργότερα. Άλλωστε είμαστε και συνάδελφοι, είστε και εσείς μέλη της Επιτροπής Αναφόρο. Είστε λοιπόν σας στο σπίτι σας, ε, είστε περιτριγισμένοι από συναδέλφους. Ελπίζω να νιώσετε άνετα. Σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Αναφορών. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχουμε να είμαστε μαζί σας σήμερα ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε σήμερα την συνεδρίασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι με ευχαριστήσατε, αλλά γιατί δεν άκουσα τη μετάφραση. Άργησε λίγο. Άργησα λίγο να φοράσω τα ακουστικά μου. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ για ό,τι είπατε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Μπορέσαμε να έρθουμε από την Σαξονία και να παρακολουθήσουμε την συνεδρίασή σας εκ μέρους της ομάδας του Τσεντεού στο Κοινοβούλιο της Σαξονίας. Θα χαρούμε πολύ σήμερα να δούμε πώς εργάζεστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά το λέω και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας και ελπίζω να νιώθετε άνετα στην Επιτροπή Αναφορών και του τουλεχθέντος. Και μετά τα σχόλια αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε το σχέδιο ημερησίας διάταξης. Ε, φαντάζομαι το έχετε μπροστά σας. Σημείο 1, πρώτο σημείο όπω πάντα, έγκριση του σχέδιου ημερησίας διάταξης. Ε, υπάρχει, κάποια, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή μπορούμε να εγκρίνουμε τη μερσιά διάταξη. Όχι. Άρα εγκρίνεται τη μερσιά διάταξη. Δεύτερο σημείο. Έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίαση τη 8η και 9η Οκτωβρίου του 2012. Σχόλια, παρατηρήσει. Όχι. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 3. Ανακοινώσει του Προέδρου τη είπα. Άρα περνάμε τώρα. Βλέπω ότι αναφέροντες έχουν αφηχθεί. Άρα μπορούμε να περάσουμε καταρχάς στις δύο πρώτες αναφορές 5 και 6. Για την 5 και την 6 έχουμε τον ίδιο αναφέροντα, αλλά μας ζητήθηκε, παρότι θα τη συζητήσουμε από κοινού, να ξεκινήσουμε από την υπαριθμόν 6. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι για το ίδιο ε, θέμα πρόκειται, λοιπόν, η αναφορά 198 του 2012 είναι από τον Ζαν Μαρί Σερβά, Γαλλική Σταγέννη και αφορά του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και την μελισσοκομεία. Παρουσία των αναφέροντο, λοιπόν. Είναι πράγματι εδώ αναφέρον ή έκανα λάθο. Και ο κύριο Σιρχά. Η αναφορά 812 τη Σίλβια Πελτράν Παγιαρή, Ισπανική Σταγέννη, εξ τη πλατφόρμα Ευρωπαία de los Conservadores del Medio σχετικά με τη θνησιμότητα των μελισσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Σαρμά, έχετε το λόγο. Θα παρουσιάσετε και τις δύο, από ό,τι κατάλαβα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί με δέχεστε ε, σήμερα στην Επιτροπή ε, μια μέρα που οι καιρικές συνθήκες πήραν το πάνω χέρι ε, στις ευρωπαϊκές μεταφορές. Θα ήθελα να αναφερθώ στα προβλήματα που προκαλούν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στη μελισσοκομεία. Βέβαια δεν είμαι ο Ζωμαρή Σελβάλε, είμαι ο Λιβιέ Μπελβάλε ε, είμαι πρόεδρος της ε, ε, Μελισσοκομικής Ομοσπονδίας, στην οποία είναι μέλη 20.000 μελισσοκόμοι. Στις 18 Νοεμβρίου του 2011 ε, έγινε ε, δεκτή, ε, μάλλον υπήρξε μια απόφαση, το, η, λεγόμενη απόφαση Βαμπλόκ, η οποία λέει ότι εάν δεν, λέει ότι δεν μπορεί ένα είδος γύρις να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε διατροφικό σκεύασμα. Δεν παρεκκλίνει ούτε το μέλι από αυτόν τον κατάλογο. οποιοδήποτε γενετικά τροποποιημένο οργανισμό χρησιμοποιούμε ε, θα πρέπει να τον επισημαίνουμε και η επισήμανση αυτή να είναι σαφή στη συσκευασία του προϊόντος. Το μέλι θεωρήθηκε ε, ε, στην αρχή ότι δεν ε, θα υφίσταται, δεν θα υπόκειται μάλλον σε αυτήν την διάταξη. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή θα πρέπει να αποτελέσει πάγια νομολογία και να αφορά και τη μελουσοκομεία οι μελισσοκόμοι ανησυχούν ε, για την επίπτωση που θα έχουν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στις μέλισσες. Απ' την άλλη πλευρά, η χρήση αυτών των οργανισμών σε 90 φορές ε, στις 100 συνδυάζονται με την χρήση ζανιοκτώνων ε, και μια γενικότερη αντιμετώπιση της γεωργίας η οποία δεν συνάδει με την μελισσοκομία, ούτε προστατεύει την υγεία των καταναλωτών η χρήση των γενετικών τροποποιημένων, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ε, μπορεί να ε, έχει ε, και σημαντικά εμπορικά και σημαντικές εμπορικές επιπτώσεις στην υγεία των κυψελών και στην ποιότητα του μελιού, πράγμα που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε αυτό το προϊόν της μελισσοκομείας. Γι' αυτό εμείς ζητούμε εφαρμογή ε, της εν λόγω απόφασης να απαγορευτεί η χρήση τροποποιημένων γενετικά οργανισμών ε, στην ε, γεωργία ε, και ε, να απαγορευθεί ε, λόγω των επιπτώσεων που έχει στην υγεία της κυψέλης και στην ποιότητα του μελιού η χρήση σε γειτονικέ περιοχές γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Δεν είμαστε μόνοι μας στο αίτημα αυτό. Οι οργανώσεις από την Γερμανία και από την Ιταλία έχουν συνεργαστεί μαζί μας και πρέπει να σας πω ότι η αίτησή μας, η αναφορά μας, συγγνώμη, είναι στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά και τώρα και στα ισπανικά. Εμείς ε, δεν έχουμε κατ' επάγγελμα ε, ε, ασχοληθεί με την δημιουργία τέτοιων αναφορών. Η δουλειά μας είναι η μελισσοκομεία, το καλό μέλι και η απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών κοντά στις κυψέλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία, τροποποίηση, η οποία όμως δεν ρυθμίζει το ζήτημα. Ε, ζητούμε ε, τροποποίηση της οδηγίας για το μέλι και το ζητούμε αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να μην ε, εμπορεύεται το μέλι το οποίο προέρχεται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν θέλουμε να γίνουμε συνένοχοι στην κατάσταση αυτή. Το, μέλι είναι προϊόν υγιεινό και είναι πρωινό αγνό. Εάν περιλαμβάνει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θέλει να βοηθήσει τους μελισσοκόμους, αλλά δεν απαγορεύει ε, την χρήση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών από όσους επιθυμούν να τους χρησιμοποιήσουμε. Θέλουμε μια πιο ριζική λύση δεν θέλουμε ε, να υπάρξει μία ψευδής ε, συμφωνία η οποία τελικά θα αποβεί προς των γεωργών. Θέλουμε ε, να προστατέψουμε και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και τις κυψέλες και το προϊόν τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ζαμαρή Μπερπά, αν είπα σωστά το όνομά σας. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ερή Κουντλέ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που ακούσαμε την άποψη των αγροτών, διότι αυτό το, το πρόβλημα με τις μέλισσες είναι πολύ σημαντικό και θα το συζητήσουμε και στο πλαίσιο της δεύτερης αναφοράς και τα ζεζανιοκτώνα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και έχουμε προσπαθήσει εδώ και πολλά χρόνια να το επιλύσουμε. Είναι ένα δύσκολο όμως πρόβλημα, δυσεπίλητο. Σε ό,τι αφορά την απόφαση του δικαστηρίου του Σεπτεμβρίου του 2011, αμέσως καταλάβαμε ότι είχε γύρει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το δικαστήριο. Το δικαστήριο όμως δεν ερμήνευσε σωστά την έννοια ε, της γύρης. Εξού προτείναμε ένα σχέδιο θεώρησε της οδηγίες για το μέλι. Στόχος μας ήταν να διευκρινιστεί ε, το καθεστώς ε, της παρουσίας γύρι στο μέλι μετά την απόφαση Μπαμπλό. Η γύρι δεν είναι ένα συστατικό το οποίο προστίθεται στο μέλι από τον μελισσοκόμο σκοπίμος. Αλλά είναι ένα φυσικό συστατικό, γιατί κατά την επικανέωση μεταφέρεται και ε, δημιουργεί, όταν δημιουργείται η κυψέλη, ε, ουσιαστικά περνάει μέσα στο μέλι. Το θέμα είναι η θεσία η επισήμανση, αν υπάρχει δηλαδή γενετικό τροποποιημένη ουσία μέσα στο μέλι. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει την Πέμπτη το θέμα αυτό με την έκθεση Γκέρλινγκ σε επιτροπή Περιβάλλοντος συγκεκριμένα. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, προβήκαμε σε ορισμένε πρωτοβουλίε, διότι πρώτα απ' όλα θέλαμε να έχουμε και μία γνωμοδότηση τη ΕΦΣΑ, τη Αρχή για την Ασφάλεια των ε, Τροφίμων, σε ό,τι αφορά τη γύρι ε, Μονσάντο 810 και τον ε, αραβόστο, τον γενικώ τροποποιημένο γιατί ξέραμε ότι δεν είχαν γίνει σχετική αξιολόγηση, υπήρχε ένα θέμα ερμηνεία για τα προϊόντα ζωική προέλευση. Όμω, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων επιβεβαίωσε ότι η γύρι αυτή που προέρχεται από το στο Μονσάντο 810 είναι το ίδιο ασφαλής με άλλες που προέρχονται από συμβατικό αραβόστο. Δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα για την ε, ανθρώπινη υγεία, ούτε και επηρεάζει ιδιαίτερα το περιβάλλον. Ζητήσαμε επίσης από την εταιρεία Μονσάντο να, κάνει, να υποβάλει ένα αίτημα ε, έγκρισης άδειας κυκλοφορίας ό,τι αφορά τη γύρω παραβώς το 810 και το Δεκέμβριο του 2012 είχαμε τη θετική απάντηση. Αυτό που απομένει λοιπόν να γίνει είναι η παράταση της ε, άδειας κυκλοφορίας Μοσάντο ε, 810 που έχει λήξει από και 4 χρόνια να ανανεωθεί, να παραταθεί. Επίσης ζητήσαμε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και τα Κοινωνικά Εργαστήρια Αναφορών να εκπονήσουν μεθόδους εξόριξης και ποσοτικοποίησης γενικώ τροποποιημένης γύρης στο μέλι, διότι υπήρχε ένα πρόβλημα μεθοδολογίας για την, ε, από, για την λήψη της ε, γύρης αυτής. Έχουμε τώρα μεθόδους ανείχνευσης στη διάθεσή μας και τα κράτη-μέλη μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να προβούν και σε απαραίτητε δοκιμές. Τελευταίο και τέταρτο σημείο. Συνύπαρξη καλλιεργιών, γενετικώς τροπημένων οργανισμών και συμβατικών καλλιεργιών σε σχέση με τη μελισσοκομεία. Ζητήσαμε από αυτό το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συνύπαρξης να μας ε, παρουσιάσει όλα αυτά τα έγγραφα συνύπαρξης ε, των ε, καλλιεργειών και τι αποστάσεις υπάρχουν μεταξύ των δύο ειδών καλλιεργειών για να μην υπάρχει επιμόλυνση από έντομα ή από τον άνεμο να μην μολυνθούν από γύρι ε, γενικώ τροπημένου οργανισμού οι συμβατικέ καλλιέργειε ή οι βιολογικέ καλλιέργειε. Και είπαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μελισσοκόμη και τη μεταφορά τη γύρι από τι μέλισσε. Δεν γνωρίζουμε ότι παραδοσιακά μία μέλισσα μπορεί να καλύψει περίπου 3 χιλιόμετρα πετώντα από την κυψέλη τη. Αυτό το έγγραφο λοιπόν του Γραφείου Συνύπαρξη πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθεί και μας δείχνει ότι η γύρη, συνολική γύρη, είναι μόνο της τάξης του 0,1% στην ποσότητα του μελιού. Να αναφέρω και κάποια από τα στοιχεία τα οποία και να τα σχολιάσω, τα στοιχεία που ανέφερα φέρω. Συγκεκριμένα, μα ζητά να μπλοκάρουμε όλου του φακέλου, ε, ό,τι σχέδιο υπάρχει ε, για τι ε, καλλιέργειε γενικώ τροποποιημένων οργανισμών που φέρουν γύρι. Μία μόνο κατηγορία αραβοσία του γενικώς τροποποιημένου ε, υπάρχει και έχει εγκριθεί το μόνο 8-10. Και μια άλλη καλλιέργεια που βέβαια δεν έχει ακόμη εγκριθεί, αλλά εκεί δεν πηγαίνουν οι μέλισσε. Και έχουμε και αραβόστο από έχουμε σόγια, βαμβάκι, πατζάρια ε, και γεώμηλα. Αλλά δεν μεταφέρουν νέκταρη γύρι, γιατί οι μέλισσε πάνε στο μέλι για να πιούν. Είτε το νερό το οποίο περιέχεται στη βάση του φύλου, είτε κάτι το οποίο ε, εξατμίζεται από τον ε, αραβόσιτο. Σε ό,τι αφορά τώρα γενετικώς τροποποιημένους, όλες μπορεί να βρίσκονται σε φυτά που φέρουν γύρι, η τοξικότητα, ενδεχόμενη τοξικότητα της γύρης για τις μέλισσες είναι κάτι το οποίο έχουμε ήδη εξετάσει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής της των Τροφίων και μάλιστα ενδελεχώς. Ζητήσαμε μάλιστα οι αξιολόγηση των ε, γάμματα να καλύπτουν τον αντίκτυπο της καλλιέργειας γάμα φόμικρων σε ε, οργανισμούς όχι στόχους ε, και συγκεκριμένα στις μέλισσες. Και συγκεκριμένα η ΕΦΣΑ καθόρισε και μια σειρά κριτηρίων για την αξιολόγηση αυτή, την επιστημονική, έτσι ώστε να προσεχθούν πάρα πολύ κίνδυνοι, ιδίως για τις μέλισσες και άλλα έντομα, αλλά κυρίως τις μέλισσες. Ο αναφέρον επίσης ζητά να είναι διαθέσιμα τα πρωτόκολλα. Αυτά τα πρωτόκολλα μελέτης γάμματα φόμικρον ήδη είναι διαθέσιμα κατόπιν ετήματος Και όλοι οι γάμματα φόμικρον έχουν αποτελέσει αντικείμενο υποβολής τέτοιου αιτήματο. Οποιοςδήποτε ζήτησε να έχει πρόσβαση στα έγγραφα για γάμματα φόμικρον έλαβε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Άρα διαθέσιμες είναι οι πληροφορίες αυτές, όχι όμως για τους πάντες, αλλά για όλους όσους έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα. Και πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή και εμείς έχουμε ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα μας υποβλήθηκε μέχρι τώρα. Δεν αρνηθήκαμε κανένα, δεν απορρίψαμε κανένα αίτημα. Απλά υπάρχουν κάποια σημεία, υπάρχουν κάποια εμπιστευτικά ε, σημεία σε ό,τι αφορά τον αριθμό των προσώπων, κάποια γενετικά χαρακτηριστικά, αλλά επαναλαμβάνω τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα και διατίθενται σε όσους τα ζητήσουν. Τέλος. Δεν βλέπω να υπάρχει ε, κάποια πρόθεση από την πλευρά της Επιτροπής ε, να σας ε, πούμε ψέματα. Είναι λίγο υπερβολικό σαν επιχείρημα αυτό. Εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι η σημασία που αποδίδουμε ως Κομισιόν στην ασφάλεια των γάμματα φόμικρων για την ε, ασφάλεια των ανθρώπων, των ζώων αλλά και για το περιβάλλον. Οι ειδικέ μας αξιολογήσεις, οι ευρωπαϊκές αξιολογήσεις θεωρούνται μεταξύ των αυστηρότερων ανά τον κόσμο και μάλιστα πολλές φορές ε, το καταγγέλουν κάποιοι, προσφεύγουν δηλαδή ε, παραγωγή ε, από χώρε που παράγουν γάμματα φόμικρο και λένε ότι είναι πάρα πολύ μακροχρόνιες οι αξιολογήσεις μας. Χώρες της Βόρειας Αμερικής σε τρει-τέσσερι μήνε ολοκληρώνεται η αξιολόγηση, εδώ πέντε-έξι χρόνια. Μάλλον σχεδόν τέσσερα-πέντε χρόνια μπορεί να διαρκεί η αξιολόγηση. Σίγουρα υπάρχουν αιτήματα για ενίσχυση και σε ό,τι αφορά την περίπτωση σύγκρουση συμφέροντων κτλ. Ναι, πράγματι, αλήθεια είναι αυτό. Εμεί όμω λέμε ότι δεν υπάρχει στον κόσμο καμιά χώρα που να είναι πιο αυστηρή η νομοθεσία για τους γάμματα φόντου. Έχουμε την πιο αυστηρή νομοθεσία. Τέλος, θα ήθελα να ολοκληρώσω με δύο σημεία. Το πρώτο είναι η καλλιέργεια γενικώ τροποποιημένου ραβοσίτου στη Γαλλία απαγορεύεται από την Εθνική Νομοθεσία. Δεν είναι κοινοτική βέβαια, αλλά απαγορεύεται η καλλιέργεια, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για τις, γα... Ε, τις γαλλικές μέλισσες. Βέβαια, ο αναφέρον λέει ότι η ένωσή του ε, δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεύτερον, για τον λόγο ακριβώς αυτό κάνουμε μια πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν ή όχι για την καλλιέργεια στο έδαφος του τέτοιων οργανισμών, αλλά με βάση κριτήρια διάφορα. Ένα από αυτά είναι η συνύπαρξη. Το κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, μέσω της έκθεσης της κυρίας Λεπάζ, ε, ήδη σε πρώτη ανάγνωση έχει συζητηθεί, έχει μπλοκαριστεί σε επίπεδο συμβουλίου από την Δανική Διπροεδρία το θέμα αυτό, αλλά βασιζόμαστε σε αυτή την πρόταση, ώστε είτε περιφερειστεί, τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίζουν σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για το κατά πόσο ε, είναι σκόπιμο ή όχι να επιτρέψουν τέτοιε καλλιέργειες. Κυρίω να απαγορεύσουν δε. Αυτό θα έλυνε και πολλά προβλήματα. Ιδίω για τους μελισσοκόμους στην προκειμένη περίπτωση. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. σα ευχαριστώ. Ε, σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον αναφέροντα. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην ασφάλεια του μελιού και των προϊόντων μελιού. Η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Αναφορών Υπήρχε μια συζήτηση για την έκθεση Σαραλίνη σχετικά με τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στο φαγητό και η θέση της ε, ΕΦΣΑ να απορρίψει την έκθεση αυτή ήταν αντικείμενο κριτικής. Υπάρχουν λοιπόν αμφιβολίες σχετικά με την ουδετερότητα της ΕΦΣΑ και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχω έρθει εδώ για να στηρίξω την αναφορά και να πιστήσω την προσοχή σας στις 6 Σεπτεμβρίου του 2011. Τότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το μέλι και άλλες πληρώματα διατροφής που περιέχουν γύρι, που προέρχεται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, δεν μπορεί να διατίθεται στην αγορά χωρίς πρώτερη έγκριση. Συμφωνώ ότι μόνο μία λύση υπάρχει εδώ για να, να προστατεύσουμε τις ε, μέλισσες. Είναι κάτι που είναι απαραίτητο και για το περιβάλλον και για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των ε, μελισσοκόμων στην Ευρώπη. Και αυτή η λύση πια είναι, ένα μορατόριο στα... στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν καλώ την Επιτροπή να ανακαλέσει την έγκριση για το τροποποιημένο καλαμπόκι MO810. και την γύρι που παράγεται από γενετικά τροποποιημένα φυτά, καθώς και να γίνει μία πλήρης έκθεση αξιολόγηση αντικτύπου και τα αποτελέσματά της να δημοσιευθούν. Τέλος, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία για το μέλι, η οποία θα συζητηθεί αυτή τη βδομάδα στην Επιτροπή ΕΝΒΗ του Κοινοβουλίου, πρέπει να γίνει μετά από μία ουδέτερη και περιεκτική μελέτη. Πιστεύω πως έχουμε συγκεντρώσει αρκετές υπογραφές ε, ως τώρα και πρέπει να κρατήσουμε το θέμα ανοιχτό μέχρι να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας πάνω στο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος στο λόγο. Ναι, βέβαια, θα σας δώσω και πάλι το λόγο. Απλά Πρέπει πρώτα να ρωτήσω αν θέλει κάποιο συνάδελφο το λόγο. Δεν βλέπω όμω να θέλει το λόγο κάποιο άλλο συνάδελφο, άρα θα σα δώσω πάλι το λόγο σε εσά, κύριε Αναφέροντα. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Από ό,τι κατάλαβα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να πει ότι για τα παράγωγα προϊόντα του μελιού ε, θα πρόκειται για μια εξαίρεση. Στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις όμως και κανονισμούς όταν μιλάμε για την ανάλυση ή την παρουσία, αν θέλετε, τροποποιημένων γονιδίων, πρέπει να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Η πρόταση της Κομισιόν είναι ουσιαστικά να παίρνει τη συνολική μάζα του μελιού ως εξαίρεση στην προκειμένη περίπτωση. Η γύρη όμω ε, του μελιού είναι αυτή η οποία περιλαμβάνει το γονίδιο, το τρόπο επιμένου στην προκειμένη περίπτωση. Άρα βλέπουμε ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ε, εξαίρεση, κάτι που δεν υπάρχει όμω για άλλα τρόφιμα. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα ε, σκαλιέργειε που ανέφερε, για τις οποίες γίνονται μελέτες για την άδεια κυκλοφορίας. Το βαμβάκι και ο αραβόστος θα αναφέρω ο Αραβόστος ε, ε, έχει γύρι. Ε, στις Κυψέλες που είναι κοντά σε καλλιέργειες έχουμε 40% των πρωτενών από εκεί και το βαμβάκι έχει και γύρι και νέκταρ. Και βλέπουμε κυρίως στην περίπτωση των Ισπανών να έχουμε πολλές επιπτώσεις. Για την περίπτωση των Ισπανών πρέπει να πω και να αποσαφηνίσω ότι πριν από δύο μέρες ο Ισπανός ε, συνάδελφος ή ε, μάλλον η μελισσοκόμη της Ισπανίας ε, καταψήφισαν την τροποποίηση της οδηγίας για το μέλι, όπως έκαναν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η Ισπανία ε, έχει αυτή τη στιγμή, ε, είναι πρώτη σε επιφάνεια καλλιεργημένη με Μονσάντο 810. Ε, δηλαδή έχει τη μεγαλύτερη επιφάνεια που είναι καλλιεργημένη με γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι και αυτοί ζητούν να μην τροποποιηθεί η οδηγία μέλη όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Χαίρομαι γιατί ακούω ότι αρχίζει αυτό να διαφαίνεται, ε, διότι ε, και όσον αφορά ε, το, τα θέματα των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων και όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς θα πρέπει να σταματήσει αυτή η συζήτηση που θα αφορά μονάχα τη σύγκρουση συμφερόντων και θα πρέπει επιτέλους να γίνουν από ανεξάρτητους οργανισμούς ανεξάρτητες και διαφανείς μελέτες έτσι ώστε αυτοί που λαμβάνουν λαμβάνουν απόφαση εν τέλει να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με τρόπο ασφαλή. Ευχαριστώ. Muy bien. Eh, vamos a ver. Λοιπόν, κύριε Τέιλορ, α, όχι, κύριε Άουκεν, Μάργαρετ, ήθελες κάτι να πεις. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να πιστεύετε ότι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι ασφαλείς και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μετά από τις εκπληκτικές διαφημίσεις της Monsanto, Δεν συζητούμε όμως αυτό. Αυτό που συζητούμε είναι ότι μέχρι τώρα ήταν απαγορευμένο και επιπλέον συζητούμε το φόρτο στους ε, μελισσοκόμους, διότι πρέπει να επισημάνουν τα προϊόντα τους εάν έχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και πιστεύω πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα υποστηρίξουμε την αποζημίωση των παραγωγών για τη ζημία που θα υποστούν στις πωλήσει μελιού επισημασμένου ότι περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Διότι ξέρετε ότι η αντιπαράθεση με τη Μονσάντο δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε απλός άνθρωπος έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, μέχρι και μέσα στην ΕΦΣΑ. Όμως, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της αποζημίωσης, το πώς θα αποζημιωθούν εάν επισημάνουν τα προϊόντα τους στην αγορά. Και πρέπει να μας ξεκαθαρίσετε, επιτροπή το πώς θα γίνει αυτό. Διότι πρέπει να έχουμε ακόμα το δικαίωμα να ε, έχουμε αυτές τις ε, επισημάνσεις. Μπορείτε κύριε της Επιτροπής ε, μέσα σε δύο-τρία λεπτά να απαντήσετε στο σχόλιο της κυρίας Σάουκεν στην ερώτησή της. Δύο λόγια μόνο κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο μέλι, βεβαίως θα πρέπει αυτό το γενετικά τροποποιημένο προϊόν να είναι να έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στην αγορά, δηλαδή να έχει αδειοδότηση. Διαφορετικά βεβαίω δεν έχουμε καμία ανοχή. Εδώ μιλάμε για τον αραβόσιτο Μονσάντο 810 ε, που σε ε, πολλές περιπτώσεις επιτρέπεται. Εάν μιλάμε για γενετικά τροποποιημένο οργανισμό που δεν έχει αδειοδότηση, το μέλι θα πρέπει να ε, καταστραφεί. Ε, απ' την άλλη πλευρά ε, πρέπει να σας πω ότι εμείς ακολουθούμε τις γνωμοδοτήσεις της ΕΦΣΑ. Εάν η ΕΦΣΑ μας πει ότι το ΑΒ ή Γ προϊόν δεν παρουσιάζει κανέναν ε, κίνδυνο είτε για την υγεία των ανθρώπων, είτε για την υγεία των ζώων, είτε για, τον περι... είτε για το περιβάλλον, τότε ε, το επιτρέπουμε. Εάν μας πει ότι παρουσιάζει ένα βαθμό κινδύνου, τότε οπωσδήποτε εμείς θα πάρουμε τα αντίστοιχα μέτρα. Με κανένα τρόπο δεν δέχομαι ότι ακολουθούμε τη Μονσάντος. Λοιπόν, υπάρχει και μία ακόμη αναφορά Νομίζω ότι ο ίδιος αναφέρουν θα μας την παρουσιάσει. Αφού ακούσουμε λοιπόν τα σχετικά με την εν λόγω αναφορά, θα ακολουθήσουμε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε και για τις δύο αναφορές. Θα το συζητήσουμε όμως μετά αυτό. Θα σας δώσω το λόγο, παρότι μια άλλη αναφέρουσα την έχει υποβάλει, κύριε Παγιάρης. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σημειώσετε εξ αρχής ότι αυτή η αναφορά δεν ξεκινά άμεσα από την δικιά μας οργάνωση, αλλά ότι η Επιτροπή Αναφορών ε, μου ζητά να υπεραμεινθώ ενός θέματος που είναι ιδιαίτερα προσφυλές στους ε, Γάλλους μιλισσοκόμους. Πρόκειται για τον αντίκτυπο φυτοφαρμακευτικών προϊόντων ε, επί των, ε, του πληθυσμού των μελισσών. Δεν γνωρίζω το ιστορικό ού, της αναφοράς αυτής, ούτε τον αριθμό των ε, υπογραφόντων, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη ε, γιατί θα αναφερθώ ε, με γενικούς όρους ε, στην αναφορά αυτή, γιατί εγώ εκπροσωπώ τους Γάλλους μελισσοκόμους. Πρόκειται για αναφορά την οποία έχει καταθέσει μια οργάνωση προστασίας περιβάλλοντος από την Ισπανία προστασία περιβάλλοντος και καταναλωτών. Ε, η αναφορά αυτή καταγγέλει τον αντίκτυπο των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων ε, επί του πληθυσμού των μελισσών. Διαπιστώνεται μια μεγάλη αύξηση της θρησιμότητας των μελισσών ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, που αποδίδεται βάσει της αναφοράς στην υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων. Ε, κυρίως δε στην ε, φιπρονίλη, την ημιδακλοπρίδη, καθώς και κάποια άλλα νεονικοτινοειδή. η, κυρίως ε, στην ε, διάρκεια της ε, ανθοφορίας των καλλιεργημένων φυτών επί των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα φυτοφάρμακα δημιουργούν πρόβλημα είτε, στις, είτε στην γύρη ε, την οποία χρησιμοποιούν ε, οι μέλισσες, είτε στα άλλα συστατικά, τα υγρά, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τον μέλι ε, οι μελισσοκόμοι και της Γαλλίας και της Ευρώπης γενικότερα αναγνωρίζουν ότι μετά από 15 με 17 χρόνια προσπαθειών των Ευρωπαίων μελισσοκόμων να ε, ε, αναφέρουν και να καταγγείλουν την μαζική θνησιμότητα των ε, μελισσών δεν καταγγέλουν λοιπόν ότι δεν έχουν καταφέρει κάτι. Στην Γαλλία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, μεγάλες αυξήσεις της θρησιμότητας του πληθυσμού των μελισσών ε, σε περιοχές που γυτνιάζουν ε, με καλλιέργειες όπου χρησιμοποιούνται εντομοκτώνα που έχουν που έχουν συστατικά όπως η φιπρινολίνη που ανέφερα προηγουμένως, η μη η ημιδακλοπρίδη, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα νεονικοτινοειδή. Θα θέλαμε να ληφθούν υπόψη είναι σοβαρά τα στοιχεία αυτά έτσι ώστε να γίνει μια σοβαρή ε, και πραγματικά ανεξάρτητη αξιολόγηση. Έχοντας ε, λάβει την προφύλαξη, ε, να, βγουν από τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων όσοι έχουν σύγκρουση συμφερόντων, διότι μετά από 17 χρόνια η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Βλέπουμε μεγάλη θνησιμότητα των μελισσών και αυτό οφείλεται στο ότι δεν ακολουθούνται σωστά τα πρωτόκολλα, διότι ε, η διεμπόρευση των προϊόντων επιτρέπεται ε, μετά από πλημελείς ελέγχους. Ζητούμε λοιπόν σε επίπεδο κρατών μελών το σύνολο των ε, εντομοκτώνων που έχουν ε, τα ενεργά συστατικά τα οποία ανέφερα προηγουμένως να ε, καταργηθούν. Υπάρχει και μία μελέτη του Μάικολ Ανρή της Ίνρα στην Γαλλία όπου, η οποία καταλήγει σε μεγάλη τοξικότητα του προϊόντος κρούζερ που χρησιμοποιείται ε, ε, ε πολύ στις ε, καλλιέργειες ακόμα και με πολύ χαμηλές δόσεις οι μέλισσες αρχίζουν να παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Εμείς πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο να αμφισβητούμε και το κατά πόσον τα στοιχεία αυτά είναι αυλαβή ακόμα και για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επομένως, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να σημειωθούν πλέον και οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται για την υγεία των καταναλωτών, ακόμα και σε πολύ χαμηλές δόσεις αυτών των προϊόντων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον εκπρόσωπο που μας ε, μίλησε και πριν, να σας ευχαριστήσω και να φέρετε και να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικότερο πρόβλημα για τις μέλησες σε, ό,τι, σε σχέση με τους χάματα φόμικρο. Το αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι είναι πιο σοβαρό αυτό το θέμα. Με τα νεονικοτινοειδή αρχίσαμε να ασχολούμαστε πριν από περίπου τρία χρόνια. Βέβαια στη Γαλλία όλα τα προβλήματα μας είχαν ήδη ε, απασχολήσει από νωρίτερα. Αλλά ήδη από το 2010 οδηγήσαμε την, ε, ενισχύσαμε την οδηγία 2010-21 που ε, ρύθμιζε την χρήση αυτών των νέων νοικοτινοειδών και δει το, την, ε, το περίβλημα σε σπόρους, στους σπόρους. Επίσης, το Μάρτιο του 2011 επανεξετάσαμε το σχήμα αξιολόγησης κινδύνων για τις μέλισσες για τη μελέτη των αυτοφαρμάκων. Ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και μάλιστα τότε δημοσιεύτηκαν και κάποια έγγραφα που θα βοηθούσαν ε, την αυστηροποίηση μεθόδου της ΕΦΣΑ για τη μελέτη των νεονικοτινοειδών και εν γέννη όλων των ζανιοκτώνων. Πράγματι, οι δημοσιεύσεις αυτές πέρυσι το 2012, γαλλικές δημοσιεύσεις, βρετανικές και γερμανικές, κινητοποίησαν ε, τον επιστημονικό κόσμο και τους μελισσοκόμους και πραγματικά προκλήθηκε ανησυχία ε, λόγω των επιστημονικών αυτών δημοσιεύσεων και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε αμέσως από την ΕΦΣΑ, την Αρχή των των Τροφίμων, να αξιολογήσει τις διάφορες αυτές μελέτες, διότι Είμαστε σε έναν ε, κόσμο πολύ ιδιαίτερο. Έχουμε ε, οξία τοξικότητα και μεγάλη θνησιμότητα για τις μέλησες λόγω των φαρμάκων, των ζυζανιοκτώνων, αλλά εδώ συγκεκριμένα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, μία τοξικότητα, υποτοξικότητα που μπορεί να μην σκοτώνει τις μέλισσες αλλά τροποποιεί τη συμπεριφορά τους. Πεθαίνουν οι μέλισσες μακριά από την κυψέλη τους και δεν, το, δεν τις ανακαλύπτουμε, δεν μπορούν να βρουν το δρόμο πίσω προς την κυψέλη. Ε, στις 7 Δεκεμβρίου δημοσίευσε ΕΦΣΑ τρεις γνωμοδοτήσεις για τις τρεις ε, ουσίες που ανέφερε και ο αναφέρον και συγκεκριμένα λέει η ΕΦΣΑ στα αγγλικά high acute risk, υψηλός οξύς κίνδυνος ε, τοξικότητας λοιπόν. Εξού σκεφτόμαστε τι δράση μπορούμε να λάβουμε και έχουμε πολλές διαφορετικές αναλλακτικές. Πώ μπορούμε τι γνωμοδοτήσει αυτέ τις επιστημονικέ να τι μετατρέψουμε σε νομοθεσία, για παράδειγμα. Ήδη μπορώ να σας πω για δύο ε, που δεν είναι σημαντικότερες. Πρώτα απ' όλα ότι θα έχουμε ενίσχυση της οδηγίας του 2010 για τους όρους χρήσης νεονικοτινοειδών και η συγκεκριμένη την προετοιμασία των σπόρων, διότι η τοξικότητα των ουσιών αυτών προέρχεται πρώτα απ' όλα και από τη σκόνη που δημιουργείται με τη φύτευση ή τη σπορά ε, αυτών των κόκκων ε, που θέλουν να προστατεύουν ουσιαστικά τα φυτά. Ένας δεύτερος άξονας είναι να ενισχύσουμε την ερευνητική δράση. Σήμερα έχουμε δύο μεγάλα ερευνητικά προγράμματα τα οποία ε, είναι το B-DOC και το b και χρηματοδοτούνται από τη ΓΑΜΑ για την έρευνα και εξετάζουν ενδεχόμενες ε, πηγές για το σύνδρομο κατάρρευσης απικιών, το CCD, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ζανιοκτώνα που μπορούν να ευθύνονται, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες ε, νόσοι, τις οποίες ε, θέλουμε να μελετήσουμε. τη βαροάση μεταξύ αυτών. Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα σύνδρομο που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά αίτια. Κάτι άλλο βέβαια είναι πολύ νωρίς για να σας πω λεπτομέρειε και θα σας εξηγήσω γιατί. Από ό,τι φαίνεται θα ληφθούν μέτρα για τη μετώπιση αυτών των τριών νέων νοικοτινοειδών. Αλλά δεν είμαι σε θέση να σας δώσω απαντήσει σήμερα. Γιατί, διότι ζητήσαμε από τις τρεις εταιρείες Time και ζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη δημοσίευση των τριών μελετών, να αντιδράσουν οι εταιρείε σε αυτές τις μελέτες. 25 του μήνα περιμένουμε τις απαντήσεις τους. Πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να ακούσουμε όλες τις πλευρές. Και τους μελισσοκόμους και τους παραγωγούς ζυζανιοκτών και τους αγρότες. Όταν λοιπόν θα έχουμε τις θέσεις των τριών αυτών, για τους μελισσοκόμους ήδη είναι γνωστή η θέση, γιατί υπήρξαν και πολλές ανακοινώσεις τύπου σχετικά. Επανέλαβε και αναφέρουν ότι ζητείται απαγόρευση των τριών αυτών ουσιών τουλάχιστον. Όταν λοιπόν θα έχουμε συλλέξει τις απόψεις και των άλλων δύο εμπλεκομένων πλευρών, Κατά πάσα πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Για τη φιπρονίλη αναμένουμε για το Μάρτιο του 2013 την γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Περιμένουμε λοιπόν την γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ και με βάση τη γνωμοδότηση αυτή θα λάβουμε τα δέοντα μέτρα σε συνάρτηση, παραλαμβάνω, και με τα συμπεράσματα των επιστημονικών μελετών για ε, τους ε, οξύς, υποξύς ή υποθανατηφόρους κινδύνους. Αυτά μπορώ να σας πω σήμερα λοιπόν και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Τέιλορ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ίσως γνωρίζουν τα μέλη, την περασμένη εβδομάδα η ΕΦΣΑ δημοσίευσε μία μελέτη για τους κινδύνους που ενδέχεται να υπάρχουν από τρία νικοτινοειδή ζυζανιοκτώνα. Δεν θα τα αναφέρω, γιατί η ονομασία είναι πολύ δύσκολη. Αλλά θα σας πω ότι η έκθεση συμπέρανε ότι μεταξύ άλλων τα ζυζανιοκτώνα αυτά αποτελούν έναν μεγάλο κίνδυνο για τις μέλισσες που τρέφονται με τη γύρη των φυτών αυτών. Επίσης, Υπάρχουν ακόμα πολλά κενά που πρέπει να συμπληρωθούν έτσι ώστε να εκτιμηθεί πλήρως ο κίνδυνος. Οι πληροφορίες για επικονιαστές εκτός των εμελισσών ήταν ελλειπής. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2012 θεωρεί ότι η χρήση ζυζανιοκτώνων έχει άμεση σχέση με τη μείωση του αριθμού των μελισσών. Και αυτό φυσικά, όπως είπε και αναγνώρισε η Επιτροπή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η οικονομική αξία της ε, μέλισσας ως επικονιαστή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εκτιμάται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί ένα μεγάλο ε, ποσοστό της οικονομικής αξίας, της οικονομικής παραγωγής. Και αυτό επηρεάζει και πολύ ε, σημαντικές οικονομικά καλλιέργειες όπως το κακάο και ο καφές. Είναι προφανές ότι εάν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι ως έχει, οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές και για το περιβάλλον και για την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια των τροφίμων. Η κατάσταση είναι επίγουσα και με βάση τις επιστημονικές ανησυχίες και τις πληροφορίες που έχουμε, θεωρούμε ότι τα ζυζανιοκτώνα αποτελούν εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο και γι' αυτό υποστηρίζω την αναφορά αυτή και υποστηρίζω την απαγόρευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των συγκεκριμένων ζυζανιοκτώνων. Η απαγόρευση έχει δεφαρμοστεί σε πολλά κράτη-μέλη και γι' αυτό καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει ένα μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση και παρακαλώ κύριε Πρόεδρε η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τέιλορ. Η κυρία Πελιάλα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. με λίγο. Γιατί νόμιζα ότι είχαν ζητήσει κι άλλοι συνάδελφοι το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, άψογα. Δεν θα επανέλθω σε αυτά που ήδη είπε ο συνάδελφος Κρίσε ε, όσον αφορά την ε, σημασία της ε, διατήρησης των μέλισσων και τον οικονομικό τους ρόλο όσον αφορά στην επικοινωνίαση των ρόλων, διότι το σημαντικό που έχουν. Έδωσε ήδη αριθμητικά στοιχεία για την οικονομία και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επικονίαση είναι ο ρόλος ο κύριος των μελισσών και επομένως έχει πάρα πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία η δουλειά τους πέρα από το οικονομικό και χρηματικό κόστος η εξαφάνιση των μελισσών θα παίξει σημαντικό ρόλο και όσον αφορά την ασφάλεια την ίδια. Ε, ε, των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το ερώτημα είναι τι μέλη γενέστε με αυτή την αναφορά. Χωρίς να επανέλθω στα στοιχεία του συναδέλφου, ε, θέλω να κάνω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα και αυτό μου φαίνεται παράδοξο ή αμφιλεγόμενο που μέχρι τώρα δεν έχουν ληφθεί καθόλου μέτρα. Δηλαδή οι πρώτες, απα... οι πρώτες ε, εκθέσεις ε, άρχισαν πριν από πολλά χρόνια, από το... μετά το 2009. Οι οικολόγοι είχαν πει επανειλημμένα ότι οι μελέτες δεν ήταν αρκετά προχωρημένες και προθυμένες όσον αφορά ε, και τη χρήση των ζανιοκτώνων και τη χρήση των ε, γενετικά τροποποιημένων ε, οργανισμών. Φτάνουμε τώρα στην αρχή του 2013 και έχουμε επιτέρους μελέτες, έχουμε τρεις επιστημονικές απόψεις οι οποίες αναγνωρίζουν την άμεση σχέση σε πολλά προϊόντα ανάμεσα στη χρήση των ζανιοκτώνων και την εθνισμότητα των μελισσών. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια διασύνδεση άμεση διασύνδεση η οποία έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Πέρα λοιπόν από την υγεία των μελισσών την ίδια, ε, παρουσιάζεται πρόβλημα ε, και κίνδυνος όσον αφορά την διατροφική αλυσίδα, άρα και την ανθρώπινη υγεία. Ερωτώ λοιπόν. Ερωτώ λοιπόν. Γιατί πρέπει να διαβουλευτούμε με το σύνολο ή να διαβουλευτείτε με το σύνολο των εμπλεκομένων. Θα μιλήσετε, δηλαδή θα ρωτήσετε τους παραγωγούς ε, ζυζανιοκτώνων και παρασιτοκτώνων εάν συμφωνούν ε, με τη μελέτη ε, θα ζητήσετε από τους, από γεωργούς ε, να πούν εάν παρά τα αποτελέσματα των μελετών, παρά την κρίση ε, της ΕΦΣΑ, αν συμφωνούν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα παρασιτοκτόνα. Ποια είναι η έννοια αυτής της διαβούλευσης. Από τη στιγμή που έχει αποφευχθεί, ε, συγγνώμη, από τη στιγμή που έχει αποδειχθεί η ίδια η άμεση σχέση ανάμεσα σε παρασιτοκτόνα εντομοκτόνα ε, και την υγεία των μελισσών. Από τη στιγμή που έχουμε εδώ πρόδειλη ε, ε, περίπτωση κινδύνου, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να διαβουλευτείτε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ποιο θα είναι το ερώτημα, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σας πω ότι ε, έχετε πράσινο φως από εμά έτσι ώστε να απογορεύσετε την χρήση προϊόντων σαν αυτά που ε, αναφέρθηκαν σήμερα και βεβαίως στηρίζω την αναφορά αυτή μέχρι ότου έχουμε ε, κοινοτική ενωσιακή οδηγία η οποία θα απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά την χρήση τέτοιων ουσιών στην Γεωργία. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο πολύ σύντομα, δύο-τρία λεπτά για να απαντήσετε σε αυτές τις ε, ερωτήσεις. Ε, και μετά θα ζητήσω και από τον ε, αναφέροντα, εάν θέλει να πάρει και αυτό το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, μία απάντηση λοιπόν στον κύριο Τέιλορ. Είναι γεγονός ότι οι τέσσερις χώρες μέλη έχουν ήδη λάβει εθνικά μέτρα εδώ και πολλά χρόνια έτσι ώστε να περιορίσουν σε, κάποιους, ε, σε κάποιες ε, ε, καλλιέργειες αυτά τα τρία, αυτές τις τρεις ουσίες, όχι όμως γενικευμένη απαγόρευση. έστω και αν αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν ε, σε παράβαση της κοινοτικής ε, νομοθεσίας. Εμείς δεν ταχτήκαμε, δεν ξεκινήσαμε διαδικασία επί παραβάση θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την ακύρωση αυτών των εθνικών νομοθεσιών, πράγμα που δεν κάναμε. Αυτό ήδη καταδεικνύει ότι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η θέση είναι μάλλον θετική όσον αφορά την ε, σταδιακή απαγόρευση αυτών των ουσιών. Απάντηση στην κυρία Ελιάς όσον αφορά το, ε, τη διαβούλευση. Κοιτάξτε, αυτή είναι η καλή ε, ε, ε, διοικητική πρακτική, δηλαδή οποτεδήποτε υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να έχει αντίκτυπο σε διάφορα σε άλλους τομείς, τότε ξεκινάμε διαβούλευση. Ξέρουμε ότι οι μέλισσες ευθύνονται ε, για 80% της επικονίασης, μάλλον για την επικονίαση 80% των ε, παραγωγμένων προϊόντων και καλλιεργιών. Έχουμε ε, ε, ε, βάσει αυτών των στοιχείων παραγωγή 17 δις τα τελευταία τρία χρόνια. Επομένως θα πρέπει να ζητήσουμε, από την άλλη πλευρά βεβαίως και η βιομηχανία δίνει δουλειά σε κόσμο και έχει μεγάλη, κατέχει μεγάλη θέση στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως θα πρέπει να συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προσπαθώντας να βρούμε μια ισορροπία και μετά την ολοκλήρωση των διεργασιών αυτών οπωσδήποτε θα κοινοποιήσουμε την θέση μας την οποία θα σας γνωστοποιήσουμε, θα μάθετε και από τον τύπο, δηλαδή από ανακοίνωθεν τύπου το οποίο θα εκδώσουμε. Ο αναφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο για το θέμα αυτό. Πολλά έχω να πω. Πρώτα απ' όλα, η γαλλική κυβέρνηση, Υπουργός Γεωργίας συγκεκριμένα, πρόσφατα πολύ ξεκάθαρα, είπε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την παραγωγή. Αυτό είναι δυνατόν για την γαλλική γεωργία αλλά και για την ευρωπαϊκή γεωργία. Δηλαδή να γίνει μια νέα γεωργική επανάσταση, αν θέλετε, προς κάτι που θα πηγαίνει πολύ περισσότερο ε, προς μια οικολογική γεωργία. Δηλαδή να έχουμε εκπεριτροπής, καλλιέργειες, πορές, ε, για να μην δημιουργούνται παράσιτα στα εδάφη και στις καλλιέργειες. Τέτοιου είδους λοιπόν γεωργία είναι ε, δυνατόν να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση που θα ευνοείται σε συστηματική προληπτική χρήση ε, των ζυζανικτών ε, με λογικό τρόπο. Εμεί μιλάμε για προληπτικά μόρια. Ξέρουμε ότι αντιβιωτικά έχουν πολύ ε, κακές επιπτώσεις και για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Σε ό,τι διαφορά τα παράστα ε, που βλέπουμε στα φυτά, ακριβώ το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Αν συσσωρεύονται ε, σύν το χρόνο όλα αυτά τα μόρια, ουσιαστικά βοηθάνε τα παράστα να αναπτύξουν μηχανισμούς ε, αντοχής. Και οι μικροοργανισμοί και έντομα μη στόχοι πλήττονται. Οι μελτοφόρες μέλισσες πλήττονται πάρα πολύ. Με σόκαρε αυτό που άκουσα, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γαλλία δεν είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο, το Συμβούλιο Επικρατεία, το Conseil d'État στη Γαλλία, κάθε χρόνο ε, τη Σιζέντα, την Μπάγερ και ε, τις άλλες εταιρείες τις ε, ε, αποφάσεις τις ακυρώνει ουσιαστικά, δεν δικαιώνει ε, τις εταιρείες. Λοιπόν, εγώ από την πλευρά μου πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έπρεπε να είχε δικαιώσει τη γαλλική κυβέρνηση εάν ήθελε να προσπίσει την απόφαση αυτή για την απόσυρση αυτών των τριών ουσιών. Σε ό,τι αφορά τώρα τις 50.000 θέσεις εργασίας της ε, αγρογεωργοχημικής βιομηχανίας, τι θα συγκρίνουμε με τις 500.000 θέσεις εργασίας που σημαίνει ε, ο μετασχηματισμός ε, ε, της γεωργίας με την οικολογική βιολογική καλλιέργεια ή 17 δις σε σχέση με 153 δις συγκεκριμένα η επιρροή των γεωργών φυτών στα, στην παγκόσμια γεωργία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Άφησε πολλά ερωτηματικά το θέμα αυτό. Ακούσαμε τι είπε και η Κομισιόν, ότι δηλαδή θεωρεί ότι είναι σοβαρό και ανησυχητικό το όλο θέμα. Ακούσαμε όλες τις πλευρές σήμερα. Σας προτείνω λοιπόν, αν συμφωνείτε, Τρία πράγματα να κάνουμε. Πρώτον, να αφήσουμε βέβαια ανοιχτέ τι αναφορέ. Το ζήτησε και ο κύριο Τέιλορ. Το δεύτερο, να έρθουμε σε επαφή με την Επιτροπή Περιβάλλοντο. Δηλαδή, στην Επιτροπή Περιβάλλοντο, στου συναδέλφου μα να του διαβιβάσουμε του σχετικού φακέλου για να εξετάσουν και αυτοί το θέμα. Και τρίτον, αν συμφωνείτε, μπορούμε να καταρτήσουμε μια προφορική ερώτηση, την οποία θα απευθύνουμε στον αρμόδιο επίτροπο εκ μέρου Επιτροπή Αναφορών για να μα διευκρινίσει ε, τη θέση της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Συμφωνείτε? Θέλετε να πείτε, να συμπληρώσετε κάτι? Όχι, ωραία. Άρα, ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτά τα δύο σημεία με τις αποφάσεις που λάβαμε και περνάμε στην υπαριθμόν 7. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες βέβαια και να περάσουμε στο σημείο 7 έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Ιταλία, 29-31 Οκτωβρίου του 2012. Έχετε την προθεσμία την κατάσταση τροπολογιών. 30 Ιανουαρίου 2013 λίγη και εγκρίνεται στις 20 Δευτέρου 2013 η εν λόγω έκθεση. Θέλει κάποιος το λόγο? Θα πάρει κάποιος το λόγο? Α, η κυρία Μέρκης, μάλιστα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη συζητήσαμε εκτενώς την διαρευνητική επίσκεψη. σε σχέση με τις αναφορές που μας ε, υποβλήθηκαν για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Ιταλία. Θα περιοριστώ αναφέροντάς σας τα συμπεράσματα και να σας αναφέρω αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα και από τότε που φύγαμε. Τα μέλη της αντιπροσωπείας γύρισαν πίσω με αρκετά κιλά χαρτιού τεκμηρίωσης που λάβαμε και από τους αναφέροντες και από τις αρμοδίες αρχές. Όποιος θέλει να συμβουλευτεί τα έγγραφα μπορεί να το κάνει. Και συμβουλευτήκαμε αυτά τα έγγραφα για να συντάξουμε την έκθεση που έχετε μπροστά σας. Η σημασία αυτής της ε, αποστολής ήταν μεγάλη για τους ανθρώπους που ανέφεραν το θέμα και για τα μέλη από την Ιταλία και για τα μέλη εκτός Ιταλίας. Επίσης, να πω ότι όλοι ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμοι και οι Ιταλικές αρχές. Στην Ιταλία υπάρχει μία μακρά παράδοση ε, αποτυχίας στην διαχείριση απορριμμάτων και έχει ζητηθεί από εμά να παρέμβουμε, ιδιαίτερα στην Νάπολη και στο Λάτσιο, στην Καμπανία, όπου το θέμα των απορριμμάτων είναι επίγουσα σημασίας. Το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και έχει γίνει έκκληση στα μέλη της αντιπροσωπείας. Αναφέρθηκε ότι η κυβέρνηση και οι τοπικές κυβερνήσεις είναι ενήμερες για το ζήτημα και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνουν οι περιοχές αυτές οι χωματερή της Ιταλίας χρειάζεται και χρειάζονται την στήριξή μας. Ωστόσο, κάποιες νέες πληροφορίες πρόκυψαν από τότε που επισκεφθήκαμε την Ιταλία. Και έχουν ως εξής. Στο Λάτσιο υπάρχει ένας ειδικός επίτροπος, όπως και παλαιότερα υπήρχε αντίστοιχα ειδικός επίτροπος στην Καμπανία. Τα μέλη της αντιπροσωπείας διατυπώνουν εξαιρετικό σκεπτικισμό για τον Επίτροπο εκείνο, αυτόν, διότι δεν ανταποκρίνεται η θέση αυτή στο πρόβλημα που υπάρχει. Υπάρχει μία μακρά ιστορία κακοδιαχείρισης και ο ειδικός αυτός επίτροπος έχει έκτακτες εξουσίες, όπως στην... και όπως έχουμε δει στην Καμπανία και στο Λάξτσιο, οι εξουσίες αυτές είναι ιδιαίτερα αντιπαραγωγικές. Πρόσφατα έμαθα ότι ο κύριος Σωτία, ο ειδικός επίτροπος στο Λάτσιο, ανέλαβε ξανά την ίδια θέση και να τονίσω με αυτό ότι εμείς η αντιπροσωπεία διατυπώνουμε έντονη κριτική για την πράξη αυτή και για τον ειδικό αυτό επίτροπο. Ιδιαίτερα όταν εκείνος έχει αναφερθεί σε σημεία που εμείς θέλαμε να αλλάξουμε. Είναι προφανές ότι η περιοχή της Καμπανίας έχει ανάγκη μόνο μία λύση. Λύση για τους χώρους ταφής απορριμμάτων. Επισκεφθήκαμε πολλές ε, περιοχές, πολλές χωματερές, οι οποίες κανονικά είχαν σχεδιαστεί ώστε να είναι προσωρινές. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι μια προσωρινή χωματερή. Αλλά σίγουρα προσωρινό δεν είναι αυτό που μένει όταν κλείσει η χωματερή. Ο Επίτροπος, ο κύριος Σωτίε, δήλωσε ότι κατά την άποψή του η έκταση της ε, γεωργίας στην περιοχή αυτή είναι ασήμαντη. Υπάρχουν 300 εκτάρια γης γύρω στην περιοχή του Λάτσιο, που είναι αποκλειστικά αφιερωμένα στην γεωργία. Και ο πληθυσμός της περιοχής δεν είχε τη δυνατότητα να υποβάλει αναφορές. Έγινε συλλογή υπογραφών, ωστόσο ο κύριος Σωτήλια έδειξε για μία ακόμη φορά ότι αγνοεί πλήρως τα παράπονα και τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής. Προφανές όμως είναι ότι το πρόβλημα αυτό επιμένει και υπάρχει, υπάρχουν αρκετά χαμηλά επίπεδα διάδρασης ανάμεσα στις αρχές και στους κατοίκους. Υπάρχουν όμως και ορισμένα ευχάριστα νέα βελτίωση της κατάστασης στην Καμπανία. Ο πληθυσμός ε, της ε, Καμπανίας, όχι μόνο στο Μόντε Ντελατάτσο, αλλά και γενικότερα, φαίνεται πως αγνοούνται πλήρως και πως αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τώρα, κάτι άλλο ανησυχητικό. Η πολιτική διαχείριση απορριμμάτων έχει δοθεί μόνο σε μία εταιρεία. Υπάρχει μία εταιρεία που έχει το μονοπόλιο λοιπόν στην ε, διαχείριση των απορριμμάτων. Πώς είναι δυνατόν σε μια τόσο μεγάλη περιοχή στην Ιταλία, σε μια τόσο σημαντική περιοχή, υπάρχει μόνο μία ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτό για εμάς είναι αδιανόητο και διατυπώνουμε την κάθετη αντίρρησή μας. Και πιστεύουμε πως αυτή η πολιτική έχει συνεισφέρει στις αρνητικές συνέπειες στην περιοχή του Λάτσιο. Επίσης, η πολιτική του μονοπωλίου έχει συνεισφέρει στην μεγάλη ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας στην περιοχή αυτή. Εμείς θεωρούμε ότι οι δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να είναι υπεράνω πάσης υποψίας και απόλυτα αντικειμενικοί. Αυτό είναι προφανές. Οι συστάσεις μας λοιπόν είναι ξεκάθαρες. Καταρχάς, αναγνωρίζουμε και επιβεβαιώνουμε τις σοβαρές κατηγορίες που διατυπώνουν οι αναφέροντες, τα σοβαρότατα ελλείμματα στη διαχείριση και των οικιακών και των βιομηχανικών απορριμμάτων στην Ιταλία. Διότι ας μην ξεχνάμε τα βιομηχανικά ελλείμματα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, Θεωρούμε πως οι πολιτικές αρχές στην Ιταλία πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν την ομαλή εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Λαμβάνουμε υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και διαπιστώνουμε δυστυχώς και άλλες παραβάσεις από πλευράς της Ιταλίας. Και θεωρούμε κατεπίγουσα σημασία η Ιταλία να αναλάβει δράση για την επίλυση του θέματος. Όπως προείπα, δεν υπάρχει επικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και τις ε, αρμόδιες αρχές στην καμπανία. Κάνουμε έκκληση λοιπόν ξανά προς τις δημόσιες αρχές να βρουν λύση ώστε να υπάρχει διαφάνεια και διάλογος με τους πολίτες. Τέλος, υπάρχουν, υπάρχουν κονδύλια τα οποία έχουν μπλοκαριστεί, κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την, ε, μια λύση στη διαχείριση των ε, απορριμμάτων. Όμως, πρώτα, οι αρμόδιες αρχές στην Ιταλία πρέπει να μας δείξουν ένα σχέδιο διαχείρισης, ένα καλό σχέδιο διαχείρισης διαπιστώσαμε μία κάποια πρόοδο, μία κάποια βελτίωση. Αργή μεν, αλλά υπαρκτή βελτίωση. Και γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει μία λύση ώστε να στηρίξει αυτές τις βελτιώσεις με τη σχετική χρηματοδότηση. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επάγρυπνοι, ιδιαίτερα στην περιοχή της Καμπανίας και στο Λάτσιο για τις εξελίξεις, πρέπει να διεξάγουμε συχνούς ελέγχους και να απαιτήσουμε τη δημοσίευση τους, τη δημοσίευση ετησίων ελέγχων και των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων. Επίσης, πρέπει να διασφαλίσουμε τον πλήρη έλεγχο των δημόσιων αρχών. και να φροντίσουμε ο νόμος να γίνεται σεβαστός από τους ιδιωτικούς φορείς που αναλαμβάνουν έργα διαχείρισης απορριμμάτων στις περιοχές αυτές. Όπως είπα, η διαχείριση απορριμμάτων αντιμετωπίζεται κυρίως από χωματερές στην Ιταλία. ο στρατός στην Ιταλία είναι παρόν στις εχωματερές και τις φυλάει. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ακριβώς ο στρατός είναι εκεί. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι μυστικά μπορεί να κρύβονται σε χώρους ταφής απορριμμάτων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητούμε επίσης την απόσυρση του στρατού από τις χωματερές αυτές, διότι αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί πάρα πολύ και μας ανησυχεί επίσης και η απόρριψη παράνομων λιμάτων και συγκεκριμένα βιομηχανικών στις χωματερές αυτές. Επίσης, παρότι στην Καπανία και το Λάτσιο έληξε ο συναγερμός, χρειαζόμαστε, πιστεύουμε, έναν νέο συναγερμό, διότι πιστεύουμε ότι οι δράσεις ε, που λαμβάνουν χώρα σχετικά με τα πορήματα είναι ανεπαρκείς και πως οι νόμοι δεν γίνονται σεβαστοί. Και πιστεύω πως είναι ξεκάθαρο ότι οι νόμοι και οι ευρωπαϊκοί και οι εθνικοί πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Διαφορετικά το τίμημα είναι βαρύ για όλους. Δυστυχώς, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον δημόσιο τομέα δεν έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις ούτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε σε επίπεδο διαχείρισης απορριμμάτων. Πιστεύουμε πως χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια στην διαχείριση των απορριμμάτων. Διαφάνεια επίσης και στις σχέσεις ανάμεσα στις περιφέρειες μεταξύ τους, διότι μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε ποιο είναι αρμόδιος γιατί. Επίσης, καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να επιληφθεί του θέματος και να δώσει διευκρινήσεις. Ήδη ανέφερα τις ανησυχίες μας για τον ειδικό αυτό επίτροπο στην Καμπανία. Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει πλέον ειδικό επίτροπος, υπάρχει αρμόδιος υπουργός στην Καμπανία, υπάρχει όμως ειδικό επίτροπος στο Λάτσιο και όπως είπα και προηγουμένως, αυτή η θέση δεν είναι σε καμία περίπτωση αρμόδια για το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Καλούμε λοιπόν να υπάρξει ένα τέλος σε αυτό το θέμα. Επίσης, πιστεύουμε ότι η αναπόθεση απορριμμάτων σε χωματερές πρέπει να σταματήσει το συντομότερο και να βρεθούν άλλες λύσεις, όπως για παράδειγμα οι εξαγωγές απορριμμάτων, έστω και ω τελευταία λύση και λύση έκτακτης ανάγκης, παρότι η οδηγία αναφέρεται σε περιφερειακές λύσεις και περιφερειακή αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων. Επίσης, πιστεύουμε ότι το μονοπόλιο αυτό στην διαχείριση των απορριμμάτων έχει πολύ βαριές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού της περιοχής. Τώρα, ας είμαστε σαφείς. Πιστεύουμε ότι η επιλογή των τοποθεσιών για τις χωματερές αυτές έγινε με πλήρως αδιαφανείς διαδικασίες, ιδιαίτερα στις περιοχές του Πιάτσιο Τελουόμο. Εμείς είμαστε αντίθετοι στην επιλογή των συγκεκριμένων τοποθεσιών. Όπως ε, προείπα, μας υπόθηκε ότι αυτές οι τοποθεσίες επιλέχθηκαν προσωρινά. Και έχουμε τις αμφιβολίες μας για την έννοια του προσωρινού. Επίσης, το θέμα της αδειοδότησης και το ποιος παίρνει αυτές τις άδειες πρέπει να υπόκειται σε συνεχούς και αυστηρούς ελέγχους. Τέλος, υπάρχει μία επιτροπή που έχει να κάνει με την διερεύνηση περιπτώσεων εγκληματιστικής δραστηριότητας στην διαχείριση απορριμμάτων. Δημιουργήθηκε τον ε, Δεκέμβρη. Το χαιρετίζουμε αυτό. Ελπίζουμε σε καλή συνεργασία και καλούμε τα μέλη της να λάβουν ενεργό δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του προβλήματος τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στην Ιταλία. Εμείς στηρίζουμε την έβρεση λύσεων, αλλά και ζητούμε από τον αρμόδιο Υπουργό να αναλάβει άμεσα δράση για τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί μέσω τη αναφορά αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρκε, λέει ο Πρόεδρο. Συμφωνώ απόλυτα πρώτα απ' όλα να πω με αυτά που είπε ο πρόεδρο πρόεδρος αντιπροσωπείας. Όλη η αντιπροσωπεία σας στηρίζει. Θα ήθελα όμως να τονίσω και κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, Ήταν καλή η επίσκεψη αυτή και θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία και τους διερμηνείς. Ήταν πάρα πολύ καλή, έκτακτη η κατάσταση και είχαμε και ένα είδος ε, εξυγχρονισμένης διερμηνίας γιατί είχαμε εξοπλισμό στην διάθεσή μας και έτσι μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Θέλω να ευχαριστήσω και την γραμματεία που φαίνεται να μαθαίνουμε στο Κοινοβούλιο πια ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και κάτι άλλο πολύ πρέπει να γνωρίζετε. Και θα συζητήσουμε και τις μελλοντικέ ερευνητικέ αποστολές. Όταν είμαστε εκεί μας αντιμετωπίζουν ως ε, τους ε, καλύτερους αν θέλετε της Ευρώπης γιατί βλέπει ο κόσμος ότι τους αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Ότι τους αντιμετωπίζουμε ως πολίτες, όχι ως αντικείμενα κακομεταχείρισης. Πολύ συχνά το βλέπουμε και το είδαμε και αυτή τη φορά. Κατοντάδες άνθρωποι να έρχονται και να μας περιμένουν. Για μία ώρα περίμεναν να μας δουν και τους ενθουσιάζει το ότι πηγαίνουν βουλευτές του Κοινοβουλίου και τους ακούνε. Δεν είναι τόσο σημαντικό τι λέμε μεταξύ μας, ε, νομίζω. Είναι τι λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Η συμμετοχή σε αντιπροσωπείες σε αυτές τις αποστολές είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι αν κάποιος θέλει και να επανεκλεγεί, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να κάνει από το να πηγαίνει σε τέτοιες αποστολές. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ καλή η ατμόσφαιρα ε, και να πω και δύο-τρία πράγματα σε σχέση με αυτά που είδαμε. Αυτό που είπατε για το ειδικό επίτροπο στο Λάτσο, πράγματι με εξέπληξε το ότι ο περιβάλλοντος πώς ήταν αρκετά καλός. Πώς ξαναδιόρισε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ε, φαίνεται να λέει ότι όλα είναι καλά, ενώ δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι περίεργο. Και σε ό,τι αφορά το κατεπήγον πράγματι, με τα απόβλητα ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και πάντα λένε κατεπήγον. Ε, αλλά τελικά τη βλέπουμε ότι μπορούν να εξαφανιστούν και όλα μπορούν να γίνουν. και τις φωτοαποτέλες που μπορούν να τις βάλουν ε, παντού μπορεί να εμφανιστούν. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά. Για το όλο θέμα με τα απόβλητα και τα απορρίμματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ιταλία, αλλά σε πολλά μέρη το αντιμετωπίζουμε. Στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στη Δανία, ξέρετε. Παρότι είμαστε οι καλύτεροι πυρομανείς, αν θέλετε, τα καίμε όλα, δεν αφήνουμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά και εκεί έχουμε πρόβλημα. Είναι όμως το ίδιο ηλίθιο να κες ή να θάβεις αυτά τα απορρίμματα που μπορεί να αποτελούν πηγή ενέργειας. Πρέπει να ανακυκλωθούν, πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτό είναι πολύ καλύτερο από αυτά που κάνουμε. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια έκθεση της Κομισιόν που λέει πόσες θέσεις εργασίας θα υπήρχαν στην Ευρώπη αν εφαρμοζόταν πραγματικά η οδηγία για τα απόβλητα και τα απορρίμματα, πάρα πολλέ θέσει εργασία θα δημιουργούνταν. Και αυτό είναι ίσω και ο ευφιέστερο τρόπο να προχωρήσουμε. Να θεωρήσουμε δηλαδή τα απορρίμματα και τα απόβλητα κάτι πολύτιμο που μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε, το ανακυκλώσουμε και το καθεξή. Οι γκάγκστερ, οι πραγματικοί, ξέρετε, δεν είναι η μαφία, είναι η πολιτική ουσιαστικά που δεν λαμβάνουν σοβαρέ υπόψη το θέμα. Πάντω θέλω να σα ευχαριστήσω για τη συνεργασία και ελπίζω να εγκριθεί έκθεση σχεδόν αυτούς όπως είναι τώρα. Πρόεδρο. ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μαγκανά, την Κομισιό. Ehm, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει ε, γνώση όλων των στοιχείων που αναφέρονται ε, στην έκθεση. Διαβάσαμε την έκθεση λοιπόν ελαμβάνομαι επίσης γνώση και των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την διάρκεια της ε, αποστολής παρατήρησης ε, που βεβαίως ε, αναφέρεται και στην κατάσταση στην περιοχή του Λάτσιο όπου τα πράγματα είναι πράγματι πολύ ρευστά όσον αφορά την περιφέρεια αυτή γνωρίζουμε ότι πρέπει να ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν αποφάσεις έτσι ώστε να μην ξεφύγει από έλεγχο η κατάσταση έτσι ώστε να μην αναγκαστούμε να έχουμε αντίστοιχη κατάσταση με την καμπάνια ε, το 2008 όσον αφορά την ίδια την ε, περιφέρεια της ε, καμπάνια όπως κατέδειξε και η αποστολή παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην καμπάνια είναι πολύ ενεργητικές ε, οι αρχές. Φαίνεται ότι έχουν μπει σε μια πολύ θετική τροχιά. Υπάρχει πλέον περιφερειακός προγραμματισμός για το θέμα αυτό. Ήδη πέρσι η περιφέρεια της ε, Καμπάνια έχει εγκρίνει ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που μελέτησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το θεώρησαν αποδεκτό. Αυτό καθόρισε και την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η οποία επισήμως ανακοίνωσε στις Ιταλικές Αρχές ε, κάποιες ειδικέ ε, κινήσεις που, πρέπει, που θα πρέπει να κάνει. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν πληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις είναι διατεθειμένη να ξεμπλοκάρει τις χρηματοδοτήσεις που είχαν μπλοκαριστεί το 2007, κυρίως όσον αφορά ε, προγράμματα τα οποία θα αφορούν τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. που ε, είναι πολύ σημαντικά σε σχέση με την ιεραρχία ε, των αποβλήτων, με την σειρά προτεραιότητας δηλαδή αντιμετώπισης των αποβλήτων. Και εδώ δεν αναφερόμαστε μονάχα στην ε, πόλη της ε, Νάπολης, αλλά και σε άλλες ε, περιοχές και κυρίως όσον αφορά την συλλογή και αποκομιδή διαλεγμένων αποβλήτων. Πρόεδρος, μου λέει γραμματή, γιατί εγώ σας είχα πει ότι μέχρι τις 30 μια ώρα θα ήταν η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών. Βλέπω όμω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη μετάφραση, όπω μου λέει η γραμματεία. Τώρα λοιπόν, 5 Φεβρουαρίου πλέον θα λήξει προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, ώστε να μπορούμε σε όλε τι γλώσσε ε, να ε, βλέπουμε τις τροπολογίες. 5 Φεβρουαρίου λοιπόν προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστήσω την κυρία Μέρκης και συνεχίζουμε με την ε, κατάθεση λοιπόν τροπολογίων και έπειτα με την έγκρισή τους αν δεν υπάρξει αλλαγή και σε αυτό, 20 Φεβρουαρίου. Στην και τώρα περνάμε στο σημείο 8, την αναφορά του κυρίου μεταρχικά DD, Βουλγαρικέ Ιθαγένειε, σχετικά με την κατασκευή ενό χώρου ταφή απορριμμάτων στην περιοχή Γιαμπόλ στη Βουλγαρία. Έχουμε μαζί μα τον αναφέροντα. Καλώ ήρθατε και έχετε το λόγο. господин председател уважаеми Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πριν λίγο άκουσα την κυρία Μέρκης να αναφέρεται στην Ιταλία. Και μου φάνηκαν γνώριμα αυτά που είπε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που έχω να παρουσιάσω την αναφορά αυτή. Ήμουν μόνιμος ε, κάτοικος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 1990 και μεγάλωσα με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστήριξα αυτές τις ε, αξίες στη Βουλγαρία κατά τα πρώτα χρόνια της ε, δημοκρατίας εκεί και τότε ήμουν αρκετά αισιόδοξο. Δυστυχώς όμως, με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι η χώρα αυτή έχει γίνει... έχει υιοθετήσει αυτά που εμείς θεωρούμε απαράδεκτα και έχουμε λάβει πολλά παράπονα για πολλά θέματα. Προσπαθούμε με διαδηλώσεις, με κοινότητας νομικές διαδικασίες και με διάφορα άλλα μέσα να κινητοποιήσουμε τις αρμόδιες αρχές και να σας πω ότι στην Βουλγαρία δεν λαμβάνεται υπόψη η υγεία των κατοίκων στο σχεδιασμό και στην χρήση χώρους ε, ταφής ε, απορριμμάτων. Ο συγκεκριμένο χώρο στο Γιάμπολ είναι πολύ επικίνδυνο και, προτι... και εμεί ε, ζητούμε να κλείσει. Η ημερομηνία που κανονικά θα έκλεινε ο Ιούλιο του 2009. Ωστόσο παραμένει μέχρι και σήμερα ενεργός και σε χρήση και έχει συγκεντρώσει έναν τεράστιο όγκο αποβλήτων. Από το 2009 μέχρι το 2012 επέκτηναν την χωματερία αυτή. Εμείς ειδοποιήσαμε τις ε, αρμόδιες αρχές για το γεγονός αυτό Και από ό,τι μαθαίνουμε τώρα συνεχίζονται τα έργα αυτά. Έπειτα, το δεύτερο αίτημα που έχουμε διατυπώσει, που έχει διατυπωθεί, είναι η κατασκευή ενός νέου χώρου ταφής απορριμμάτων στο Γιάμπολ. Θα επιθυμούσαμε αυτή η οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων να εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή και να γίνει μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Προσπαθήσαμε να συναντηθούμε με τον ε, κύριο Ράσμουσεν της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συναντηθήκαμε, το καταφέραμε και του εξηγήσαμε τα προβλήματα. Με συγχωρείτε, μάλλον όχι, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συναντηθούμε με εκείνον. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε επίσης και με τον κύριο Κράμπλης, ο οποίος είναι επικεφαλής του τομέα περιφερειακής ανάπτυξης, για να υπάρξει μια συνεργασία και με τις ε, αρχές της Βουλγαρίας. Αυτό που λάβαμε ως απάντηση όμως είναι ότι η απόφαση για, την, τον ορισμό χώρων ταφής ε, αποβλήτων είναι απόφαση των, ε, της βουλγαρικής κυβέρνησης. Όμως οι, οδηγοί, οι ευρωπαϊκές οδηγίες ε, για τους χώρους αυτούς προβλέπουν το ακριβώς αντίθετο. Τα άρθρα 6 έως 15. Έπειτα υπάρχει και άλλη ευρωπαϊκή οδηγία για τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις αντικτύπου όσον αφορά τα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα, άρθρο 2, παράγραφος 3. Επίσης, οι πρακτικές της Βουλγαρίας παραβιάζουν τις, τα άρθρα 5, 6 και 8 της Ευρωπαϊκής ε, Οδηγίας για προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, παραβιάζει και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την δημιουργία πλαισίου για τις ε, δράσεις όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και τον υδροφορό ορίζοντα και παραβιάζει και ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικούς με την περιφερειακή ανάπτυξη. και διεθνείς συμβάσεις, συμβάσεις για την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα και συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πολιτική της Βουλγαρίας επίσης παραβιάζει και την εθνική νομοθεσία. ιδιαίτερα νόμους για διαχείριση αποβλήτων, ε, νόμους για τα ύδατα, για την πολιτιστική κληρονομιά, για την πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες. και νομοθεσία για την επιλογή χώρων επεξεργασίας αποβλήτων και για τις μελέτες, υγειονομικές μελέτες σε αστικά κέντρα. Η κατάσταση στο Γιάνμπολ έχει περιγραφεί εκτενώς στην αναφορά μας. Καταρχάς, δεν έχει γίνει ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και η άδεια που έχει ο χώρος αυτός δεν ανταποκρίνεται στις διαστάσεις του. Η άδεια είναι για μικρότερους ε, χώρους ταφής απορριμμάτων. Έπειτα, η επιλογή της τοποθεσίας της χωματερής αυτής δεν είναι εναρμονισμένη με την εθνική νομοθεσία. Μετά, χωρητικότητα της τοποθεσίας αυτής. Η χωρητικότητα δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επίσης δεν έχει διεξαχθεί καμία ανάλυση όσον αφορά τις ποσότητες και την εμορφολογία των αποβλήτων που καταλήγουν στο Γιάμπολ από τις πέντε διαφορετικές ε, αστικές περιοχές. Έπειτα, δεν έχουν γίνει μελέτες στην, ε, όσον αφορά την ποιότητα του νερού και τις διαρροές στον υδροφόρο ορίζοντα. Μετά, έχει δοθεί παράνομα άδεια σε δεύτερη, σε δεύτερη εταιρεία και δεν έχει γίνει η ανάλογη περιβαλλοντική μελέτη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο επίσης έχει λάβει αποφάσεις οι οποίες έχουν ακυρωθεί από το δικαστήριο ως παράνομες. Και αυτή τη στιγμή το θέμα δεν έχει λήξει δικαστικά. Επίσης, να σας πω ότι η περίπτωση του Γιάμπολ με αφορά και προσωπικά. Το πατρικό μου σπίτι βρίσκεται κοντά στην περιοχή αυτή. Και κοντά και στην περιοχή που έχει προταθεί ως επέκταση. Ε, εμείς ε, έχουμε απευθυνθεί και στην, ε, στο Δικαστήριο Δημιουργίου Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Σήμερα απευθύνομαι ενώπιον σας σαν εκπρόσωπος του κινήματος για το περιβάλλον. Έχουμε 2.350 ε, υπογραφές ε, άλλων ε, πολιτών συγγνώμη, της περιοχής που αντιτίθενται στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων στον χώρο υγειονομικής ταφής του Γιάμπολ. Επίσης και πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη την στήριξη της ε, συστημικής αντιμετώπισης ε, των ε, χώρων υγειονομικής ταφής. Έχουμε έρθει σε επαφή ε, και με τις αρχές διαχείρισης των αποβλήτων. Και ζητούμε επίσης και από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος να μας δώσει όλα τα στοιχεία ε, τα οποία αφορούν τα, τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτού του ε, έργου. Να μας δώσει λοιπόν όλα τα έγγραφα τα οποία είναι υποστηρικτικά αυτού του έργου. Εμείς ζητήσαμε ε, και από το Ευρωπαϊκό Λογικό Κόμμα, στην οικογένεια του οποίου ανήκει ε, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, να δει το θέμα αυτό. Η Βουλγαρία, οι πολίτες της Βουλγαρίας ζητούν βεβαίως και χρειάζονται την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των περιοχών τους. Αλλά αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλήγει στη δημιουργία υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τις επόμενες γενναίες. Για λόγους οικονομίας χρόνου θα ήθελα απλώς να πω ότι έχουμε λεπτομερή φάκελο που ακολουθεί την ε, αναφορά μας. Σας προσκαλούμε λοιπόν να επισκεφθείτε επιτόπου την θέση του Γιάμπολ και όταν θα έρθετε στο Γιάμπολ να μην μιλήσετε μονάχα με τις αρχές, να μιλήσετε και με εμάς. Εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα έχει παρακαλώ το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω βουλγαρικά καθότι είναι εδώ βούλγαρος ε, αναφέρον ε, και υπάρχουν και βουλγαροί ε, βουλευτές. Θα απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Δεν θέλω να επαναλάβω το νομικό πλαίσιο. Απλά θα σας ε, κάνω μια ιστορική αναδρομή από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά τον φυστάμενο χιτά στο Γιάμπολ, που λειτουργεί κατά παράβαση της ε, οδηγίας 31, υπάρχει διαδικασία παραβάση, δυνάμει του άρθρου 258, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα τέλη Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε μια αιτιολογημένη γνώμη προς την Βουλγαρία και αυτό ήταν το δεύτερο ε, τελευταίο και τελευταίο στάδιο της προκαταρκτικής περίοδου. Η Βουλγαρία ε, εφόσον δεν ε, αντιδράσει, θα προσφύγουμε στο δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή, τη δημιουργία ενός νέου χιτά στο χώρο αυτό αλλά και σε γειτονικού δήμους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές μέσω του λεγόμενου EU Pilot, ενός πιλωτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έρχεται σε επαφή με διοικητικούς φορείς των κρατών μελών πριν ξεκινήσει διαδικασίε επί παραβάση δυνάμει του άρθρου 258. Στι αρχέ του τρέχοντο μηνό λοιπόν, λάβαμε την απάντηση από τη Βουλγαρία σε όλες μας ε, τις ερωτήσεις σχέση με αυτή τη νέα χωματερή και σε σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μας εξηγήθηκαν οι τεχνικές πτυχές ε, και η δυναμικότητα αυτού του νέου χώρου, η χωρητικότητά του. Η απάντηση που λάβαμε μας λέει ότι έχει παγώσει το πρόγραμμα διότι υπήρχε μια επενδυτική πρόταση που αποσύρθηκε και αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή αναστολή των όλων εργασιών. Μια πρόταση πάντως δεν υπάρχει. Αυτή λοιπόν σήμερα είναι η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να προβαίνει σε οποιαδήποτε δέουσα ενέργεια σε σχέση με την ε, κατασκευή νέων χιτά που συγχρονατοδοτούνται μέσω περιβαλλοντικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πληρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις. Θα πρέπει να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συζητήσουμε τις εκκρεμείς υποθέσεις, γιατί πρώτα πρέπει να αποφανθούν τα εθνικά δικαστήρια. Ολοκληρώνοντας, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει άμεσα στην επιλογή τοποθεσιών για τη δημιουργία νέων χιτά. Βέβαια, θα πρέπει να τηρείται σίγουρα η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να επαληθεύσουμε. Πρόεδρος, ποιος θέλει το λόγο, κύριε Άουκεν. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον αναφέροντα και κατάλαβα καλά. Τα έχετε καταφέρει πάρα πολύ καλά, είστε πολύ αποτελεσματικός, διότι αν, αν έχει ε, διακοπεί το project αυτό, ε, πρέπει να συγχαρούμε γι' αυτό, φαντάζομαι. Δύο-τρία σχόλια. Πρώτα απ' όλα, αν είναι αλήθεια ότι κάποιος προσπάθησε να ξεφορτωθεί, αν θέλετε, την ε, μελέτη αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, δεν θα είναι, αν σας το πω, η Βουλγαρία η μόνη χώρα. Δεύτερον, και επειδή ήμουν πρόεδρος μιας διερευνητικής επιστολής στη Βουλγαρία πέρυσι, πρέπει να πω ότι η Βουλγαρία σίγουρα έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις, για να το θέσω έτσι. Και τα απόβλητα είναι μία των προκλήσεων αυτών. Και δεν είναι και πολύ ξεκάθαρη η σχέση μεταξύ εργολάβων, αρχών. Πραγματικά κάποιες φορές με σόκαρε ε, η διαπίστωση ότι είναι πολύ συνδεδεμένη Είμαι μένε με τους δε. Και τελικά δεν καταλάβαινα ποιος διαπραγματεύεται, οι αρχές ή οι αργολάβοι. Δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο πάντα αυτό. Πολλές φορές έχω διαπιστώσει για τη Βουλγαρία ότι υπάρχει όμως μια κοινότητα των πολιτών πάρα πολύ δραστήρια και πάρα πολύ ικανή. Και το λέω αυτό στραφών και προς τους αναφέροντες που είναι εδώ σήμερα, αλλά αυτό είναι και ένα μήνυμα. Βέβαια το γνωρίζει σίγουρα η Κομισιόν αλλά και για τις αρχές της Βουλγαρίας είναι ένα μήνυμα. Προσέξτε, προσέξτε, διότι υπάρχει ε, αυτή η κοινωνία των πολιτών που έχει πολύ μεγάλη αξία, όταν δηλαδή ο κόσμος ε, καταλαβαίνει και νιώθει ότι πρέπει να συμμετέχει, να κάνει αναφορές, να γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, να ασχολείται με το τι γίνεται. Άρα Δράτω με τις ευκαιρίες για να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι πρέπει να στηρίζουμε εμείς από την Επιτροπή Αναφορών την Κοινωνία των Πολιτών για να κρατήσει την ίδια στάση. Και βέβαια όταν ε, εργάζονται τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να τα αφήσουν να επιτελέσουν το έργο τους, αλλά είναι ταυτόχρονα και πολύ καλό όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση, να παρακολουθούμε τα πράγματα. Τέλος να πω ότι η σύμβαση που είναι δανέζικη είναι μια σύμβαση που πάντοτε την υποστηρίζουμε και είναι δύσκολο, ξέρετε, γιατί δημιουργήθηκε για να δώσει την κοινότητα των πολιτών κάποια βασικά εργαλεία για να διαδραματίσουν το ρόλο τους οι πολίτες και πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες. Ε, μιλάμε για την παλιά σήμαση λοιπόν και για την οδηγία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Λοιπόν, εγώ λέω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να μην ανοιχτεί. Okay. Κύριε Γιώτοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα βουλγαρικά γιατί εδώ έχουμε διάφορους ε, ε, βουλγάρους φίλους στην αντιπροσωπεία. Κοιτάξτε, αυτή είναι πέτ ευρωπαϊκή διεκτήβη. Από ό,τι έχουμε ακούσει, υπάρχουν πέντε παραβιάσεις ευρωπαϊκών οδηγιών και εθνικής νομοθεσίας. Και αυτό που ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι οι πληροφορίες από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας ε, είναι ότι οι επενδύσεις έχουν παγώσει ή έχουν αποσυρθεί. Ωστόσο, μας δόθηκαν κάποιες εγγύησεις ότι οι επόμενες επενδύσεις δεν θα παραβιάζουν ευρωπαϊκή εθνική νομοθεσία και τα project θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται παραβιάζοντας όλες τις ε, περιβαλλοντικές ε, προδιαγραφές, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων. Και πιστεύω ότι καλό θα ήταν να παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, πριν από τη δίκη σχετικά με το κλείσιμο της επροτινόμενης χωματερής να δούμε, και να δούμε πώς θα διεξαχθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες για το νέο προτινόμενο χώρο. Προτείνω λοιπόν η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, φίλους από τη Βουλγαρία. Γιατί πιστεύω επίσης ότι και για τη Μάργαρετ και για εσάς είναι <clears throat> σαν τεζαβού μετά την επίσκεψη το 2011 στη Σόφια. Είδατε ότι τα προβλήματα παραμένουν και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ίδια. και ότι οι βλάβες και οι ζημιέ προ το περιβάλλον έρχονται και από την ε, πλευρά της ε, κυβέρνηση και αυτό με σοκάρει και εμένα και τη Μάργαρετ και άλλους. Και μας όταν η αρμόδια υπουργό ε, Περιβάλλοντος μας είπε πόσο μεγάλη είναι η δέσμευση τη βουλγαρικής κυβέρνηση να εφαρμόσει και να υιοθετήσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πόσο σοβαρή, σοβαρά έχουν πάρει το θέμα της εφαρμογής και των ε, περιβαλλοντικών μελετών. Και τι βλέπουμε τώρα. Αυτό που βλέπουμε τώρα στην περίπτωση του Γιάμπολ και στην αναφορά αυτή που υποβλήθηκε από την ΜΚΟ που βρίσκεται σήμερα μαζί μας, τι δείχνει. Δείχνει πρώτον φτωχή εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και είναι προφανές αυτό. Είναι οφθαλμοφανές. Και το αποδέχεται μέχρι και η κυβέρνηση στη Βουλγαρία. Δύο, φτωχή εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις περιβαλλοντικές μελέτες και μονόπλευρη. Εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να σταματήσει την διαδικασία αξιολόγησης του project και τρίτον, είναι γνωστό το θέμα με τις ε, καθυστερήσεις και τις περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη καλούνται από την Επιτροπή και τους αναφέροντες να δώσουν μια απάντηση στις ε, θεμητές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι σαν τις ε... ελληνικές καλένδες. Υπάρχουν κατηγορίες για παραβιάσεις, για παραβάσεις, για διαφθορά, μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων και των πηγών οι οποίες είναι ζωτική σημασία για τις κοινότητες της περιοχής αυτής. Τέλος, ε, πώς να το πω για να μην προσβάλλω κανέναν. Πώς να αναφερθώ για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους, στις ε, ΜΚΟ τις αγνοούν πλήρως. Και όχι μόνο αυτό, δεν έχουν και πρόσβαση σε επίσημες πληροφορίες, δημόσιες πληροφορίες σχετικά με ένα project. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στην περίπτωση της Βουλγαρίας γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Τώρα, ας δούμε την περίπτωση Σφότο, που μοιάζει πάρα πολύ με την περίπτωση του Γιάμπολ. Ο χώρος αυτός βρίσκονταν κοντά στη Σόφια και αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι, συνεχι... ότι μιλάμε για μια συνεχιζόμενη παραβίαση ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων στη Βουλγαρία. Δεν μπορούμε να το ωρεοποιήσουμε. Αυτό είναι. Και το 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα, χρηματοδο... και θα ψηφίσει επίσης ειδικέ ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή project χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η δημιουργία νέων κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. και να ζητήσουν από τα κράτη-μέλη να απαντήσουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς και να δούμε πώς μετά από το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δαπανίσει άσκοπα περαιτέρω κονδύλια για έργα τα οποία είναι σε αντίθεση, σε απόλυτη αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρο, κύριο Στινάρου. Κύριο Στινάρου, ζητήσατε το λόγο, αλλά να είστε σύντομος, παρακαλώ. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Όσον αφορά τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλες παρόμοιες οργανώσεις να πω το εξής. Δεν έχουμε πληροφορηθεί για το τι έχει συμβεί. Και όσον αφορά την απόσυρση των ε, επενδύσεων, να πω ότι αυτή η πληροφορία δεν είναι απόλυτα αληθής. Χάρη στην, στον οργανισμό μας, επενδύσαμε πάρα πολύ χρόνο για να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την εξέλιξη αυτού του project. Συγκεντρώσαμε όλες τις ε, παραβιάσεις της νομοθεσίας και μετά όταν τις υποβάλαμε αποσύρθηκε η επένδυση εν μέρη. τώρα Μα αναφέρεται ότι ήδη είχε υπογραφεί σύμφαση με την ε, τοπική κυβέρνηση του Γιάμπολ για την κατασκευή τη χωματερή χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη και χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Και δεν ούτε καν παραδέχτηκαν πως ζήτησαν συγχρηματοδότηση και ούτε πως συζήτησαν με την ε, κυβέρνηση του Γιάμπολ για ένα νέο χώρο ταφής. Ευχαριστώ πολύ. Άρα θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Θα παραμείνει ανοιχτή, παραλαμβάνω, αναφορά. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη. Πρέπει να στείλουμε μια επιστολή στη βουλγαρική κυβέρνηση για να απαντήσουν σε σχέση με τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν εδώ. Mm. Συμφωνείτε να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα περνάμε στην αναφορά 9. Αναφορά 212 του 2008 του Ιωάννη Παπαδόπουλου Βελγική Ιφαγέννη σχετικά με την κατασκευή χώρων υγειονομική τάφη απορριμμάτων στην Ελλάδα. Κυρίε Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Αναφορών, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που για τρίτη φορά ε, με δέχεστε εδώ. Να σας πω εξ αρχής ότι ε, μόνο σήμερα το μεσημέρι έμαθα ότι έπρεπε να εμφανιστώ ενώπιό σας. Δεν ξέρω ε, για ποιο σκοτεινό λόγο έφτασε τόσο αργοπορημένη η πρόσκλησή μου. Να σας πω επίσης ότι από το Φεβρουάριο του 2008 ισχύει η αναφορά μου ε, και λόγω των πολλών καθυστερήσεων τελικά έλαβε χώρα αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή που σας ανήγγειλα το 2008. Πλέον έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και επιστημονικώς αποδεικνύεται αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή. Στην 3η Νοεμβρίου του 2009 είχα αναφερθεί ε, στην, ε, ε, στον χιτά του Καρβουναρίου, στην Θεσπρωτεία και στην Κέρκυρα στη Λευκήμη. δεν θα μιλήσω πολύ για αυτά τα θέματα αυτά, γιατί τώρα στη Λευκήμη, ας πούμε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί ε, ε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής ε, οι οποίες θεμελιώθηκαν και πάνω στο πτώμα μιας νεαρής γυναίκας που σκότωσαν τα ΜΑΤ και αυτή τη στιγμή φυλάσσεται αλλά δεν λειτουργεί διότι οι πολίτες της Λευκήμης ήταν πάρα πολύ δραστήριοι στις διαμαρτυρίες τους και κανείς δεν τολμάει να θέσει σε λειτουργία την, τον χιτά της Λευκήμης. Το καρβουνάρι είναι μια άλλη ιστορία. Στο Καρβουνάρι λοιπόν λειτουργεί ο ΧΙΤΑ. Σας είχα δείξει τότε πώς ε, είχε ξεπεραστεί η βούληση του κόσμου και θα επανέλθω σε ένα σημείο μόνο. Σε αυτήν την άλλη, τον άλλο χιτά της ε, θες πρωτείας την Κορίνθιανη και θα μιλήσω πριν για αυτήν. Ε, πρόκειται για έναν χιτά ο οποίος το 1999 δημιουργήθηκε από, με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999 που δεν λειτουργήσε όμως ποτέ. Στην Κορίτιανη λοιπόν σε ένα έγγραφο που έχω εδώ μπροστά μου. Το είχα κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα ότι δεν λειτουργεί αυτός ο χώρος ε, ταφής. Ζήτησε λοιπόν τα ρέστα από την, Ευρωπαϊκή, από την ελληνική κυβέρνηση ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη σειρά της η, ελληνική κυβέρνηση άρχισε, ε, έθεσε σε λειτουργία αυτόν τον χιτά της Κορίτιανης χωρίς όμως άδεια λειτουργίας. Άδεια λειτουργίας πήρε μονάχα το 2011. Το γράφει εδώ, τον Μάρτιο του 2011. Είχε κατασκευαστεί από το 1999, δεν είχε ε, χρησιμοποιηθεί, δεν είχε λειτουργήσει ποτέ και μετά από όλη αυτή την κατάσταση που δημιούργησε το καρβουνάρι πήρανε άδεια και για το 2011. Στην ουσία δηλαδή κατασκευάστηκε μονάχα για να ε, ε, πάρουν οι αρμόδιοι τα χρήματα και όχι για να υπάρχει ένα πραγματικός, ένας πραγματικός ε, χιτά. Αυτή τη στιγμή πώς είναι η κατάσταση, έχει γεμίσει τόσο πολύ ο χιτά που έχει κλείσει πλέον και όλα τα απορρίμματα τα οποία θα έπρεπε, των οποίων η αποκομιδή θα έπρεπε να γίνεται στον χιτά της Κορίτιανης, τελικά φτάνουν στο καρβουνάρι. Επανήλθε, λοιπόν για μια δεύτερη παρουσίαση τον Δεκέμβριο του 2011, 20 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα του 2011 και εντωμεταξύ είχα ε, ευρία ανταλλαγή επιστολών με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει τη διαδικασία του 2009 40-43, την οποία μετά ολοκλήρωσαν, έκλεισαν. Στις 20 Δεκεμβρίου του 2011 δεν υπάρχει Έλληνας βουλευτής αλλά πάντως την προηγουμένη την 19η Δεκεμβρίου δηλαδή, αυτός ο κύριος που θα σας δείξω τώρα μόλις τον βρω, αυτός ο κύριος, τον οποίο ενδεχομένως γνωρίζετε, είναι ο διαβόητος κύριος Κωνσταντίνου, παλαιός ε, τέος ε, Υπουργός Οικονομικών και τότε ε, Υπουργός Περιβάλλοντος. Ε, ε, ο τότε λοιπόν υπουργό τη 19η Δεκεμβρίου είχε μαζέψει όλους τους βουλευτές για να τους μιλήσει για, τη, για τον χιτά ε, στο Καρβουνάρι, στη Λευκήμη, καθώς επίσης και για τον άλλο χιτά στην Πελοπόννησο. Ήταν και βουλευτέ εδώ. Η κυρία Παλιαδέλη μάλιστα του είπε ότι θα πρέπει να κλείσει αυτό ο χιτά. Ε, σας δείχνω τη φωτογραφία αυτή γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπακοσταντίνου ε, διώκεται για παραχάραξη και, και χρήση πλαστογραφημένων εγγράφων ε, σχετικά με την λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ. Ε, γιατί αυτός, ο κύριος Παπακοσταντίνου δηλαδή, χωρίς καμία ντροπή, ε, παραχάραξε, τροποποίησε και αλλίωσε τη λίστα Λαγκάρντ. Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Και σας το λέω το ευτυχώς, διότι ε, τώρα πλέον η, ε, ε, ε δημόσιοι υπάλληλοι της Ελλάδος έχουν απελευθερωθεί από αυτό το ζυγό που είχαν μέχρι τώρα. Αισθάνονται ελεύθεροι πλέον να κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Πρέπει να σας πω ότι παλιότερα, λόγω της τεράστιας, της τρομερής πολιτικής πίεσης που υφίσταντο, ε, να κρύβουν πράγματα. Ε, και ε, γι' αυτό ακριβώς ε, μπορούμε τώρα να επανέλθουμε στο Καρβουνάρι και εδώ έχω και ένα έγγραφο 40 σελίδων. εκπλήσω με σας λέω πραγματικά με το έγγραφο αυτό. Γιατί μ, υπάρχουν εδώ άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, οι οποίοι δεν έχουν καμία γνώση γεωλογίας ή γνώση ε, ε υπογείων υδάτων κτλ. Εγώ, εγώ, ο Αδαής, τα είχα αναφέρει όλα αυτά και τα είχα πει, τα είχα στείλει και τα είχα κοινοποιήσει τα προβλήματα αυτά ε, στους ε, περιβαλλοντολόγους που χρησιμοποιούσε το Υπουργείο. Είπα ότι υπήρχαν προβλήματα ε, αποβλήτων επικινδύνων. Είπα ότι υπήρχαν αποβλήματα, συγγνώμη, προβλήματα διαφυγής διασταλαζών των υγρών. Είχα πει ένα σωρό πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως στις διάφορες επιστολές της υπεραμείνθηκε της ελληνικής κυβέρνησης. Παραθέτω, 31 Μαρτίου του 2010. Ε, αναφέρετε επίσης στην ε, ε μήνυσή σας ε, ότι ε, υπάρχει μεγάλη, υπάρχει σειρά, σειρά διατάξεων οι οποίες παραβιάζονται. Όμως ε, σας λέγω ότι υπάρχει ε, διαρκής έλεγχος της φρουρούμενης ε, χωματερής σχετικά με το ποια είναι τα απορρίμματα, τα, οποία, τα απόβλητα τα οποία εισάγονται. Υπάρχει έλεγχος, στήριση μητρώου κτλ. Ο χώρος προστατεύεται και φυλάσσεται κτλ. Τον εισερχόμενων με εκφόρτωση φορτίου στην είσοδο του χιτά έρχεται σε αντίθεση με τον περιβαλλοντικό όρο Δέλτα 2.1, Δέλτα της 25 σχετικής απόφασης ε, ε, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και με το άρθρο 3, παράρτημα 1, κεφάλαιο, κεφάλαιο, κεφάλαιο. Ça, c'est un des exemples. Alors, on me dit, dans, dans cette réponse que la στην απάντηση λοιπόν ε, που μας δίνει η Επιτροπή ε, λέει ότι στο σεβασμό, ε, όσον αφορά τον σεβασμό των αρχών αναφέρεται επίσης Il doit être noté que tous les lixivias sont gardés dans le site. Ε, ε, ότι τα επικίνδυνα απορρίμματα ε, φυλάσσονται, ελέγχονται, διαλέγονται κτλ. κτλ. Και ότι υπάρχει στεγανοποίηση και επομένως συλλογή και διαχείριση των διασταλαζών των υγρών. Διαρροής στραγγισμάτων. Η μελέτη, κατασκευή και παραλαβή των λειτουργικών έργων υποδομών γεωτρήσεις και η μη έγκαιρη λήψη μέτρων για την επίτευξη του σκοπού κατασκευής έλεγχος διαρροής στραγγισμάτων θέτει ζητήματα ορθότητας των στοιχείων μελέτης και κατασκευής τους καθώς και νομιμότητας της παραλαβής αυτών. Μπορώ να συνεχίσω. Απαντώ λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους λέω δεν ισχύει αυτό που μου λέτε αγαπητοί κύριοι και στις 11 Ιουνίου του 10 ε, μου λένε ότι όχι δεν ισχύουν αυτά που λέω μου λένε ας πούμε. Δεν πρόκειται να σας τα διαβάσω όλα γιατί είναι πολλές σελίδε. Μου λένε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όταν παραπονιέμαι ότι υπάρχει ένας αγωγός ε, ο οποίος βγάζει τα νερά από την χιτά. Κοιτάξτε, εγώ έλεγα ότι στην Ελλάδα ε, όλες οι, όλοι οι χιτά χτίζονται πάνω σε ε, και γιατί στην ουσία το πρόβλημα είναι η διαχείριση των στραγγιδίων και ότι στην ουσία η τελική ε, ε, ε, εν τέλει αυτά τα υγρά χύνονται είτε σε ποτάμια είτε σε, στην ακτή, είτε στη θάλασσα. Εγώ είχα διατυπώσει μια υπόθεση που μετά όμως επιβεβαιώθηκε γιατί οι ίδιοι οι ελεκτές περιβάλλοντος το είχαν πει και στο Καρβουνάρι μάλιστα είπαμε ότι υπάρχει ένας αγωγός ο οποίος, ο οποίος ρίχνει τα, τα στραγγίδια στην, ε, ε, στον παρακείμενο ποταμό. Και μάλιστα ε, είναι αυτός ο ποταμός ο οποίος αποτελεί την μυθική πύλη εισόδου στην, στον Άδη. η λοιπόν. Εδώ αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμία ε, διαφυγή ε, υγρού και ότι έχει μονοθεί με τσιμέντο μάλιστα ο ογός αυτός ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί μονάχα στη διάρκεια των ε, έργων κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής. Τι μου λένε λοιπόν εδώ. Rappelle que la lettre de la Commission est 11 juin 11 Ιουνίου του 10, ε, έτσι έγινε, μου γράψανε αυτήν την, ε, την επιστολή, αλλά ε, μετά από μερικούς μήνες αναφέρεται ότι... ...από PVC διατομής ΦΥ 250 με απόλυξη σε υδατόρεμα σε απόσταση 40 μέτρων περίπου κατάντι του φρεατίου συλλογής στραγγισμάτων. Το υδατόρεμα έχει μικρή ροή ενός λίτρου ώρα περίπου. Τα ρέοντα υγρά ήταν ελαφρώς κουρόχρωμα χωρίς ιδιαίτερη οσμή. Στο σημείο υπήρχε ανεπτυγμένη ομονοητή και πολιτή χλωρίδα. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο λειτουργία, ο σωλήνα τοποθετήθηκε κατά, κατά την κατασκευή του έργου. Με την ανάληψη τη λειτουργία από τον ανάδοχο, διαπιστώθηκε η ροή πιθανών στραγγισμάτων στο εν λόγω σημείο, Μάρτιο 2012. Ο ανάδοχο λειτουργία ενημέρωσε εγγράφο του αρμόδιου φορεί και με πρωτοβουλία του τοποθέτησε το πόμα. Παρά την τοποθέτηση του πόματο, η ροή του υγρού στο υδατόρεμα βγαίνει αυξομοιούμενη ανάλογα με τι καιρικέ συνθήκε. Ζητήθηκε και προσκομίθηκε η σχετική αλληλογραφία με του φορεί. Ensuite, que font les Τι κάνουν μετά, οι ε, ε, ελεγκτές παίρνουν το υγρό και το αναλύουν. Προκύπτουν υψηλέ τιμέ COD, BOD5 και αγωγημότητας ε, η τιμή αυτή, και μάλιστα λέει... αυτή θεωρείται υπερβολικά υψηλή και αναφέρεται με επιφύλαξη. Donc, Επομένως αυτή η μόλυνση έχει αξία τόσο ψηλή που, ε, ε αμφιβάλλουν αν πραγματικά ισχύει αυτή η τιμή. Πασμένα και γι' αυτό υποβαθμισμένα νερά. Δεδομένη τη ανυπαρξία σημειακών πηγών ρήπανση ανθρωπογενού προέλευση στην εγγύη του έργου περιοχή, τεκμέρεται ότι η επιβάρυνση των υδάτων προκαλείται από τη λειτουργία του χιτά. και έχω εδώ και μία σειρά από άλλα στοιχεία, δεν μπορώ όμως να ξοδέψω το χρόνο σας ε, αναλύοντάς σας τα. Όμως να σας πω ότι το Μάρτιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου είπε σε μία επιστολή της, πάρα πολύ απλά, να το βρω μόνο δύο λεπτά, τον Ιούλιο μάλλον, τον Ιούλιο,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 δεν μπόρεσα να βάλω τα χαρτιά μου σε μια σειρά γιατί σήμερα το μεσημέρι μου είπαν ότι πρέπει να έρθω. Εν πάση περιπτώσει μου έλεγε ότι δεν είναι ε, ορθό και χρήσιμο να ε, συνεχιστεί αυτή η αναφορά και η μήνυση διότι ε, συμμορφούται αυτή, αυτή, αυτός ο χιτά με όλες τις αρχές. Λοιπόν, όμως με έκπληξή μου βλέπω ένα έγγραφο στην, ε, στο, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής όπου αναφέρεται σε μια τελική εκδοχή της Δευτέρας Ιουλίου του 2012 και αναφέρεται ας πούμε στην Ελλάδα για τη διαχείριση αποβλήπων όπου λέει ότι η, ε, η Ελλάδα δίνει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μονάχα ένας από τους ε, χιτά συμμορφούται με τις οδηγίες. Δηλαδή η ίδια η Επιτροπή που τον, τον Δεκέμβριο μου έλεγε ότι όλα είναι εξαιρετικά, στην τελική της δική της αναφορά ε, λέει ότι ε, από όλου του χιτά που έχουν χρηματοδοτηθεί στην ε, Ελλάδα, μονάχα ένας, να, να, υποθέσω ότι είναι στο καρβουνάρι, λειτουργεί συμμορφούμενο με όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2011 είχα δώσει κι άλλο ένα έγγραφο Όλοι, όλος ο προγραμματισμός ε, της διαχείρισης αποβλήτων στην ε, ε, Ελλάδα είναι λάθος, είναι εσφαλμένη και μάλιστα σε μία συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή ο κύριος Κρεμλίσε το είχε αναγνωρίσει αλλά από την άλλη πλευρά είχε εγκρίνει την χρηματοδότηση χιτά τύπου γραμματικού. Αυτά που σας είπα για το καρβουνάρι ισχύει και για το ελληνικό, για την άλλη μεγάλη, ε, τον άλλο μεγάλο χιτά και για το γραμματικό και για την κορίτιανη. Στην κορίτιανη μάλιστα είδατε ε, τι συνέβη. Ακριβώς λόγω του ότι εμείς ήρθαμε εδώ και διαμαρτυρηθήκαμε και γνωστοποιήθηκε το θέμα, αρχίσαν να λειτουργούν τον χιτά στην κορίτιανη γρήγορα γρήγορα έτσι ώστε να μην ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Θα σας ξαναδώσω όμως ε, ε, και το έγγραφο της ε, μελέτης των, της πραγματογνωμοσύνης των εμπειρογνωμόνων της, των περιβαλλοντικών εμπειρογνωμόνων που επιτέλους μπορέσανε να ξεφύγουν, να ελευθερωθούν από την σοβαρή πολιτική πίεση λόγω της κρίσης και να μπορέσουν να πούνε την αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στην Κομισιόν. Βέβαια δεν ήξεραν και αυτοί τα προβλήματα που είχατε και εσείς. Ζητώ συγγνώμη που δεν ενημερωθήκατε νωρί. Ελπίζω να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να μην ενημερωθείτε την τελευταία στιγμή. Να σας ευχαριστήσω πάντως κύριε Παπαδόπουλε και να δώσω το λόγο στον κύριο Κουνινιώτη, αν το είπα καλά το όνομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι πληροφορίες που θα δώσω στην Επιτροπή σας ελπίζω τουλάχιστον ότι θα ικανοποιήσουν και τον αναφέροντα. Ο αναφέρον ξεκαθάρισε ένα ερώτημα που είχα ότι μιλούσε για τους δύο αρχικούς χιτά που ανέφερε και όχι γενικώ τις χωματερές στην Ελλάδα. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση για την Κορίτιανή και να πω ότι ε, είναι αληθεί οι ισχυρισμοί του αναφέροντος και έχουμε κίνηση στα δικαστήρια σε παραβάση βασιζόμενη ιδίω στην απουσία άδεια. Οι ελληνικέ αρχέ εξέδωσαν την άδεια, ενημερώσαμε τον αναφέροντα που ήταν και καταγγέλων τότε και με τη βάση αυτή έκλεισε τότε η καταγγελία αυτή και διαδικασία παραβάση. Από ό,τι κατάλαβα σήμερα, υπάρχουν κάποια ακόμη δεδομένα τα οποία δεν έχουμε εμεί στη διάθεσή μα και θα ήμουν ευγνώμων ε, μέσω τη Επιτροπή σα, αν αναφέρουν μπορεί να μα τα διαβιβάσει, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε τα ε, δέοντα μέτρα για την ε, λόγο χωματερή. Και κλείω την παρένθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά του δύο χιτά τη Λευκήμη, πρώτον, όπω είπα, αναφέρουν δεν, δεν έχουμε εξελίξεις εκεί, έχει πλέον ολοκληρωθεί το project, αλλά δεν λειτουργεί. Δεν θα επανέλθω σε αυτό που είχε πει η Κομισιόν στην τελευταία ανακοίνωση, δηλαδή ότι υπήρχε μια μελέτη ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πληρούσε τις διαταξεις του οδικές 2011-92 τώρα και σε ό,τι αφορά την οδηγία 9931 για τα απόρριτα και τις 2008-98 ε, ε, την οδηγία πλαίσιο. Πληρούνταν λοιπόν η διατάξα. Πρέπει να δούμε βέβαια αν η Λευκίνη θα λειτουργήσει για να δούμε τελικά αν πληρούνται όλες αυτές οι απαιτήσει. Κάτι όμως πολύ πιο σημαντικό τώρα σε σχέση με το καρβουνάρι. Είχαμε ενημερώσει την Επιτροπή σας στην τελευταία μας ανακοίνωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε βάσει των στοιχείων που μας χορήγησε ο αναφέρον, νομίζω το Μάρτιο του 2012, να ανοίξουμε ένα φάκελο EU Pilot και να απευθύνουμε ερωτήματα σε ελληνικές αρχές. Αυτό φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρει τον αναφέροντα, όλο ιδιαίτερο με βάση τι απαντήσει των ελληνικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε άμεσα και άνοιξε ένα νέο φάκελο, ε, διαδικασία επί παραβάση 2012-2208 είναι η αναφορά, το reference number, λόγω των προβλημάτων που διαπιστώσαν και κατά την επιθεώρηση, τα ανέφερε και ο αναφέρ. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε για τον κατάλογο, παραδείγματο χάρη σε υδατόρευμα που χύνονται από έναν αγωγό λίματα και διαχείριση αερίου είναι έναν άλλο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω όμω ότι την 5η στι 24 Ιανουαρίου θα ε, συζητηθεί ε, στο Σώμα των Επιτρόπων και θα πρέπει να αποφασιστεί κατά πόσο πρέπει να στείλουμε προειδοποίηση ε, στην Ελλάδα για την συγκεκριμένη αυτή υπόθεση. Βέβαια θα σας στηρίσουμε ενήμερους μέσω ανακοίνωσης, πρόσθετης ανακοίνωσης. Τώρα, θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια σημεία που ανέφερε ο αναφέρον στην παρουσίασή του. Για παράδειγμα και συγκεκριμένα να μιλήσω πάλι για αυτό τον αγωγό, για αυτό το σωλήνα. Όπως λέει και ο αναφέρον, η Κομισιόν τότε, νομίζω το 2011 ήταν, μπορεί και νωρίτερα, είχε έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, αναφέροντας ε, τα στοιχεία τα σχετικά με σχέδια διαβιβάσεων αναφέρουν και οι ελληνικέ αρχέ μα είχαν διαβεβαιώσει ότι ναι, δεν υπήρχε αυτό ο αγωγό, αλλά είχε τσιμεντωθεί. Άρα ήταν ε, κλειστό, δεν λειτουργούσε. Όπω όμω ε, δηλώνουν και οι επιθεωρητέ, φαίνεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα, όχι μόνο από πλευρά παραβίαση τη περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά είναι και θέμα ενδεχόμενη παραβίαση ε, των ε, υποχρεώσεων που έχει το ελληνικό κράτο απέναντι στο, στην Επιτροπή. Δηλαδή, αν σκοπίμω και εσκεμμένα ψεύδεται προ την Κομισιόν ένα κράτο μέλο, αυτό είναι σημαντικό, είναι σοβαρό. Και λυπούμε που δεν έχει Κομισιόν αυτή τη στιγμή δυνατότητα να ε, πάει επί τόπου να επιθεωρήσει. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Βέβαια, εμπιστευόμαστε τις ελληνικές αρχές. Για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω ότι ο αναφέρον πάρα πολύ σωστά και δικαιολογημένα διερωτάται γιατί μόνο τώρα αντιδράσαμε στους κομισιόν. Ξέραμε από τη φάση του σχεδιασμού ότι υπήρχαν προβλήματα. Δεν θέλω να επανέλθω σε όλα όσα έχουμε πει και στις προηγούμενες ανακοινώσεις μας ε, εδώ στην Επιτροπή σας, αλλά να θα αναφέρω το εξής. Η κατάσταση ήταν τέτοια που πριν να αρχίσει να λειτουργεί ΧΙΤΑ, μετά το σχεδιασμό και τη μελέτη πριν τη λειτουργία όμως, τη θέση λειτουργία, θέλαμε να δούμε την συμβατότητα του, της, ε, της περιβαλλοντικής οδηγίας για τις περιβαλλοντικές πτώσεις. Θέλαμε να δούμε αν τηρούνται οι διατάξεις οδηγίας 92-2011. Και είδαμε ότι ναι, τηρούνταν οι σχετικέ διατάξει, άρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά τι οδηγίε για τα απόβλητα, αφού δεν είχε αρχίσει να λειτουργεί οχητά και οι ελληνικέ αρχέ μπορούσαν ακόμη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ε, σύμμορφη λειτουργία. Από τη στιγμή όμω, που ξεκίνησε η φάση λειτουργία, η Κομισιόν άμεσα επαλήθευσε βάσει και τη έκθεση τη επιθεώρηση που σας έστειλε ο αναφέρον, αν η λειτουργία αυτή ήταν πράγματι σύμμορφη. Και από ό,τι φαίνεται, και είναι σαφές αυτό, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή και γι' αυτό το τον επιτρόπο, την Πέμπτη, όπως σας είπα, θα λάβει απόφαση για το κατά πόσον πρέπει να στείλει προειδοποίηση στην Ελλάδα ή όχι. Και για να ολοκληρώσω, θα σχολιάσω και την οδηγία EIA για τη μελέτη περιβατικών επιπτώσεων. Η οδηγία αυτή σήμερα όπως έχει, έχει κενά. Εξού και η Κομισιόν προτείνει μια νέα οδηγία για να προσφέρουμε περισσότερες εγγύησεις και να αποφύγουμε έτσι ή να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Και είδα στην μερσιά διάταξη μάλιστα ότι η Επιτροπή σας ε, θα αγγίψει ε, αύριο συγκεκριμένα σε αυτό το ζήτημα. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, για να δούμε, για να δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ε, σύντροφος που θέλει να λάβει το λόγο. Εγώ πριν δώσω το λόγο στον αναφέροντα, θέλω να πω το εξή. Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ο αναφέρον έκανε μια καταγγελία που κατά την άποψή μου, αλλά νομίζω και κατά την άποψη όλων των ε, βουλευτών που ε, άκουσαν, ε, είναι κάτι που πρέπει να το καταγγείλουμε ή τέλο πάντων να το ρωτήσουμε. Και εγώ ρωτώ απευθεία εσά. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχύει, ξέρετε ότι με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιήθηκαν αγωγοί που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, μάλλον δόθηκαν χρήματα και δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ για την κατασκευή αυτού του αγωγού. Excusez-moi, Αν αληθεύει ότι μια χωματερή μάλλον, που είχε δημιουργηθεί στην Ελλάδα με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Έχετε πληροφορίες ή όχι. Αν αναφέρει στην Κορίτιανη δεν έχω πληροφορίες. Αν χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια, αποδεσμεύτηκαν κονδύλια και δεν λειτουργεί αυτή η χειροκομματερή, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το δούμε με τις αρχές. Ε, Δυστυχώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Τρία-τέσσερα λεπτά έχουμε μόνο στη διάθεσή μας. Αν μπορείτε λοιπόν να είστε πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Και να απαντήσετε. Ναι, αυτό που λέτε πραγματικά ισχύει, δηλαδή δεν λειτουργήσε ποτέ αυτή, αυτός ο χιτά. Ε, ε, δεν έχω τώρα τη διαφάνεια, αλλά στη διαφάνεια είχα ε, το ποσό το οποίο πληρώθηκε από το Β, από το δεύτερο κοινοτικό ε, πλαίσιο στήριξης, από το Ταμείο Συνοχής. Ε, χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, αλλά χρησιμοποιήθηκε, άρχισε να λειτουργεί δηλαδή, μονάχα όταν εγώ ξεκίνησα όλη αυτή τη διαδικασία με τις καταγγελίες και τα λοιπά. Και πρέπει να σας πω ότι ο αρχιτέκτονας αυτής της χιτά που ζούσε τότε στην ε, περιοχή και είχε κάνει πολλά έργα ε, με, το, τα χρήματα του Ταμείου Συνοχής ε, πριν από το 2008 βέβαια και ο οποίος τώρα είναι υπεύθυνος για τον δημοσιονομικό έλεγχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είχε εκλεγεί πλέον βουλευτής. Είναι πραγματικά λυπηρό ε, το ότι γεγονός ότι στο Καρβουνάρι έπρεπε να περιμένουμε να έχουμε μόλυνση των υπογείων υδάτων, μόλυνση ε, λοιπόν της περιοχής, μόλυνση του ε, παρακείμενου ποταμού έτσι ώστε ε, να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες. Είναι τρομερό το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι δίνουν τα χρήματα ή χρηματοδοτούσες αρχές εν προκειμένου η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, δεν ε, ε, μπορούν να ελέγξουν εκ των προτέρων και θα σας πω ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε ούτε τον κύριο Φούχτελ ούτε τον κύριο Ράιχεμπαχ για να μας ελέγξουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι θέλουν το καλό της Ελλάδας. Σε όλες τις πολιτικές οικογένειες υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προστατεύσουν το καλό της Ελλάδας όχι με αυτόν τον τρόπο όμως με τον σωστό τρόπο. Πρόεδρος. Επομένως, προτείνω να αφήσουμε ανοιχτή είναι την αναφορά. Και να σας πω ότι στα τέλη του Μαΐου η Επιτροπή Αναφορών θα επισκεφθεί την Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα έχουμε τότε και την ευκαιρία, αν συμφωνείτε κι εσείς βέβαια, να επισκεφθούμε αυτόν τον χιτά ε, και να συμπεριλάβουμε λοιπόν στο ταξίδι μας ε, τις, ε, τους χιτά αυτούς, τους, οι οποίοι έχουν αποτελέσει αντικείμενο κάποιων αναφορών. Ναι, δεν σας είχα δει, θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Η κυρία πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπρόσωπους της Επιτροπής να θέσουν στη διάθεσή μας τις σχετικές πληροφορίες και θα ήθελα επίση να ρωτήσω μέχρι πότε μπορούμε να τις περιμένουμε. Ευχαριστώ. Ε, κύριε εκπρόσωπο της Επιτροπής, εννοείται ε, δόκιμες πληροφορίες, αναφέρετε το, την ε, ε, συνέχεια που θα δοθεί στο ε, θέμα αυτό, κοιτάξτε, η Γενική Διεύθυνση πλέον και φαντάζομαι ότι εν ευθέτω χρόνο ή εν πάση μόλις έχει την πρότασή της ε, θα σας την διαβιβάσει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ρωτώ για την οικονομική κατάσταση, τις λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση. Όσον αφορά αυτό το σημείο θα έρθω σε επαφή με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Ρέγγιο. Δεν είναι θέμα περιβαλλοντικό αυτό καθεαυτό. Η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο έχει όλα τα στοιχεία. Δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα πότε θα μας τα δώσουν. Θα προσπαθήσω πάντως ακόμα αύριο να σας τα στείλω. Ε, πότε ακριβώς, μέχρι πότε. Δεν μπορώ να απαντήσω εξ ονόματός τους. Εγώ θα κάνω το αίτημα όπως σας είπα αύριο. Ο, μόλις μου στείλουν τις ε, πληροφορίες θα σας τις ε, στείλω κι εγώ με τη σειρά μου. Πρόκειται για πληροφορίες τις οποίες θεωρητικώς έχουν ήδη στη διάθεσή τους, επομένως δεν θα είναι δύσκολο. Πρόεδρος, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και μετά να ακολουθήσετε και το αίτημα της συναδέλφου και να στείλετε όσο γίνεται πιο γρήγορα τις πληροφορίες, κύριε Βίλα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή Αύριο, αν μπορέσουμε να αλλάξουμε τα σημεία 7 και 14, το σημείο που αναφέρεται στη Ρουμανία, διότι τις ημέρες αυτές μου ανακοινώθηκε μία άλλη αναφορά σχετικά με ένα ταμιευτήριο στην Ρουμανία. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα. Έπειτα, να σας ε, κάνω έκκληση, επίγουσα έκκληση. Να ασχοληθούμε με την αναφορά αυτή σχετικά, ε, σε συνδυασμό με την μετρόσοφυλα. Χωρίς εγνωμοδότηση δεν μπορούμε να ε, συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Και η αναφορά αυτή έχει υποβληθεί από την επιστημονική κοινότητα, από κάποιον που έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ. Είμαστε, θα γίνουμε γελοί στα μάτια τη επιστημονική κοινότητα αν το καθυστερήσουμε. Το σημειώνουμε λοιπόν. Θα στήσω από τη γραμματεία το στομότερο δυνατό να σα δώσω αυτά τα στοιχεία, ιδίω ό,τι αφορά το 47, αν άκουσα καλά τον κύριο Βίλαντ. Και πριν αύριο λάβουμε απόφαση, θα ενημερώσω τον κύριο Βίλαντ σε σχέση με το αίτημά του Κύριε Βίλαντ, όμως μας προλάβατε, γιατί δεν είχαμε λήξει με το θέμα αυτό. Μας μένει μια αναφορά και με αυτήν θα ολοκληρώσουμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα πριν από τις συνεδρίες των συντονιστών και συγκεκριμένα είναι η 10 ε, ε, αρχικά LAG Ισπανικής Ιθαγένειας αναφέρον ε, για την μόλις του ποταμού Δουέρου με μη επεξεργασμένα λίματα. Κατά παράβαση της οδηγίας 91 κάθετος 271 κάθετος ΙΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Η αναφορά 922-2011. Ο κύριος Χωσέφαλο Μαρτίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ισπανικά για να επικοινωνήσω και με εσά αλλά και με τα μέλη τη Επιτροπή σα. Η λόγω αναφορά η οποία απεστάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαβιβάστηκε σε εμά μιλάει για ενδεχόμενο μη τήρηση οδηγία για τα αστικά λίμματα και εξηγεί μια περίπτωση όπου τα λίμματα τα οποία προέρχονται από ένα μικρό οικισμό 200 και περίπου κάτοικοι φαίνεται ότι αυτά τα λήματα πέφτουν στον ποταμό Δουέρο χωρίς επεξεργασία προηγούμενη. Στα έγγραφα τα οποία σας διαβιβάσαμε βλέπουμε ότι οι Ισπανικές αρχές αυτή τη στιγμή θεωρούν και έχουν υπόψη τους ότι πρόκειται για παρανομία ε, σε ό,τι αφορά την ε, Ισπανική Ενωμητάξη και κατά την άποψη της Κομισιόν θεωρούμε ότι ενδεχομένως αυτό συνιστά και παράβαση του άρθρο 7 της οδηγίας για τα λύματα. Είναι περίεργο ε, που παρότι αναγνωρίζουν λοιπόν ότι δεν υπάρχει παράβαση, το αναγνωρίζουν οι Ισπανικές Αρχές, δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο για την ε, διόρθωση της κατάστασης. Επομένως, σε κάθε περίπτωση ε, η Κομισιόν δεν μπορεί να κάνει και πολλά παραπάνω για να υποχρεώσει τις Ισπανικές Αρχές να προχωρήσουν και γιατί υπάρχει απόφαση ή μάλλον υπάρχει ένα διοικητικό πόρισμα που δείχνει ότι υπάρχει παράβαση και δεύτερον γιατί λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος του οικισμού αυτού, σας είπα πρόκειται για 200 κατοίκους και επειδή υπάρχει ενδεχόμενο παράβασης ε, του άρθρου 7, η Κομισιόν δεν μπορεί ακόμη να ξεκινήσει να αναλύει ε, την τήρηση μη του άρθρου αυτού και πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα κεντρωνόμαστε από πλευράς Κομισιόν ε, στο να εξασφαλίσουμε την τήρηση των ε, βασικών διατάξεων της οδηγίας αυτής ε, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη συλλογή λιμάτων, την επεξεργασία τους και κυρίως για τους μεγάλους οικισμούς, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό το, με, το, μέσο που χρησιμοποιούμε είναι η λεγόμενη οριζόντια διαδικασία για κάθε κράτος μέλος, όπου όλα τα αστικά κέντρα που υποτίθεται ότι παραβιάζουν ε, την νομοθεσία ε, εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να σας πω ότι και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές ε, έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την επίλυση τέτοιου είδου προβλημάτων διότι απαιτείται, όπως είπα, μια σε βάθος γνώση Τη ε, της κατάστασης του περιβάλλοντος και θα πρέπει κανείς να γνωρίζει επίσης και τα διοικητικά ε, και νομικά ε, συστήματα και στοιχεία που συνιστούν αυτή την παράβιαση οδηγία. Θα Θέλω να σα πω εν τέλει ότι η Κομισιόν δραστηριοποιείται έντονα για το θέμα αυτό. Έχει ανοιχτέ πολλέ νομικέ διαδικασίε σε βάρο πολλών κρατών μελών και δι πρώτη πρώτης κρατών. Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει ήδη καταδικαστεί για παράληψη σε ό,τι αφορά την τήρηση των άρθρων 3 και 4 ε, και έχει προσφύγει Κομισιόν κατά τη Ισπανίας στο δικαστήριο γιατί δεν τηρούνται διατάξεις για την επεξεργασία βάσης των υδάτων. Έχουμε στείλει και προειδοποίηση στην Ισπανία σε ό,τι αφορά τους μικρούς λεγόμενους οικισμούς, δηλαδή μεταξύ 2 και 7.000 κατοίκων. Επειδή οι Ισπανικές αρχές ε, αντιλαμβάνονται ότι ενδεχομένως ε, υπάρχει παράβαση ε, της οδηγίας και επειδή είναι η κατάσταση ως είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω στο παρόν στάδιο. Πρόεδρος, θέλει κάποιος το λόγο? Όχι. Αν κανείς δεν θέλει το λόγο, τότε μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά. Από ότι μου είπαν και επειδή δεν έχουν απαντήσει οι Ισπανικές αρχές, θα μπορούσαμε και για να τους ενημερώσουμε ενδεχομένω ε, να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ενημερώσει. Είναι περίεργο. Ε, μήπως πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η αναφορά. Να τους ρωτήσετε γιατί δεν απάντησαν, γιατί δεν απάντησαν σε αυτή την αναφορά. <coughs> Αν συμφωνείτε.